Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ στις θέσεις σας. Ξεκινούμε τη συνεδρίαση, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να βεβαιωθώ ότι η διάταξη προς πρώτη να με σας βρίσκει σύμφωνος. Η κυρία Τζόρτζεβα, αντιπρόεδρος, έχει επιβεβαιώσει την αύξηση εδώ, ε, σήμερα στις 11.30 για την παρουσίαση νέων πρωτοβουλειών ε, για την αντιμετώπιση των κατεπηγουσών αναγκών. Άρα πρέπει να αλλάξει η ημερήσια διάταξη ως εξής. Η ημερήσια διάταξη για το πρωί. θα δει πρώτα την παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της αποστολής μας στην Τουρκία πριν από ένα μήνα. Μετά το σημείο 8 της κυρίας Καρδιά Ζαμπάλ, Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική, συνέπειες για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια. Μετά θα δούμε το 4 ενημέρωση σχετικά με τον τριμερή διάλογο της 14 Μαρτίου 2016. Το πέντε πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις στο πλαίσιο του Προπολογισμού για το 2016 και το 2017. Και τελευταίο για το πρωινό, το νούμερο 6 παρουσίασε από την Επίτροπο κυρία Τζόρτζεβα για τις νέες πρωτοβουλίες σχετικά με την παροχή στήριξη έκτακτη ανάγκη εντό τη Ένωση. και αυτό κατόπιν για να απαντήσω σε παρατήρηση του κυρίου Φερνάντες ε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας των συντονιστών. Το απόγευμα. Η κυρία Τρίπελ με το σημείο 9 της τωρινής ημερής διάταξης. έλεγχος του Μητρώου και τη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων αναβάλλονται για τις 4 ε, και 10. Οι ψηφοφορίες αρχίζουν στις 4.40. Ε, Το σημείο του κύριου Ταραντ θα πάει για μετά τις ψηφοφορίες, δηλαδή κάπου στις 5 ε, ε, για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου ΔΕ η συζήτηση θα γίνει και κλεισμένων των θυρών καθώς πρόκειται για ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια και καθώς στην προηγούμενη συνεδρίαση παρουσία του Γενικού Γραμματέα και του Αντιπροέδρου κ. Βίλαντ υπήρξαν ζητήματα καθώς ορισμένα ερωτήματα δεν μπόρεσαν να ε, απαντηθούν διεξοδικά. Δεδομένου ότι γινόταν μέσω του διαδικτύου ή μετάδοση του τη συνεδριάσεως ε, και άρα μπορεί οι απαντήσεις που μας δίνονταν να έφταναν σε ότα ενδεχομένως ακόμη και τρομοκρατών. Ε, γι' αυτό λοιπόν σήμερα έχουμε και κλεισμένων των θυρών τη συνεδρίαση. Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 9 με 12.30 γίνεται συνεδρίαση μεικτή με την Οικονομική Επιτροπή στην ε, αίθουσα Γιάννα 1 6Q2. Συντονιστές οι συντονιστές αποφασίζουν 15 Ιουνίου να γίνει συνεδρίαση ακροάσεων με τις επιτροπές ΑΦΕΤ, ΝΤΕΒΕ και ΛΥΜΠΕ για τις δημοσιονομικές συνέπειες της μεταναστευτικής κρίσης. Για δε τις αποστολές μας, μια αποστολή που είχαμε για το Λίβανο και την Ιορδανία αποφασίζουμε να διεξαχθεί από 16 Μαΐου έως 19, Δευτέρα με 5η Μαΐου. 16 με 19 Μαΐου. Συντονιστές. Για έκθεση πρωτοβουλίας για την κοινή γεωργική πολιτική. Ποια είναι τα μέσα που μπορούν να μειώσουν την πτυτικότητα των τιμών στις, γεωργικές, ε, στις αγορές γεωργικών προϊόντων. Οι Άλντε, φιλελεύθεροι να λαμβάνουν, με τον κύριο Αλή. Ευρωπαϊκή Ένωση Άμυνας, Αμυντική Ένωση. Έκθεση του άρθρου 53. Ο υποφαινόμενος και πρόεδρός σας. ΑΚΕ, Παύλα Ευρωπαϊκή Ένωση, δύο τελείες, ποιες σχέσεις μέχρι το 2020, ε, οι φιλελεύθεροι δημοκράτες η Ευρώπη των Ελευθεριών και των Δημοκρατιών. Μακροοικονομική ε, ενίσχυση στην Τινησία αποστέλλεται επιστολή στην Επιτροπή Ίντα. Επίσης, οι συντονιστές έλαβαν την απόφαση να αποστείλουν επιστολή στην Επιτροπή σε σχέση με το ζήτημα των revolving doors, δηλαδή της ανάληψης από παλαιούς επιτρόπους νέων δραστηριοτήτων, συναφών ενδεχομένως με την παλαιά τους εντολή και ζητήματα ύψους αμοιβών και ενδεχομένων συγκρούσεων συμφερόντων. Ο κύριος Ταράντ που τέρος εκφράσει ανησυχίε του το θέμα αυτό. Μας έχει υποστείλει τις επιστολές που απίφθηνε ο ίδιος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακόμη δεν έχουν λάβει απάντηση προκειμένου να διευκρινιστεί η κατάσταση. Αυτά είχα να σας ενημερώσω. Τα πρακτικά σχέδια πρακτικών της των συνεδριάσεων 27 Οκτωβρίου 2015, 27 Ιανουαρίου 2016, 15 Φεβρουαρίου 2016, 18 Φεβρουαρίου 2016, 23 Φεβρουαρίου 2016. Έχετε λάβει, έχετε παρατηρήσεις. Εάν όχι. Εγκρίνονται. Και τώρα. Αποστολή. Τουρκία. Εξ ονόματος της ε, ομάδας των συναδέλφων της Επιτροπής μας που επισκέφθη την ε, Τουρκία με την αποστολή αυτή, θέλω να σας δώσω τις πληροφορίες μας, πληροφορίες που συλλέξαμε, αλλά και εμπειρίες μας από την αποστολή αυτή, καθώς και μηνύματα και συμπεράσματα που πιστεύουμε πως είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε. Πρόκειται για μια αποστολή που συνιστά σημαντική συμβολή στις τρέχουσες εργασίες της Επιτροπής των Προϋπολογισμών. Σημειώνω δε ότι επιστρέφοντας από την αποστολή αυτή είδαμε την εξέλιξη και άλλων ε, γεγονότων με τραγικές πολλές φορές διαστάσεις. Μια μετρική εκεχηρία στη Συρία έχει ανακηρυχθεί, έχει διακηρυχθεί. Μάλιστα ενημερωθήκαμε το μεταξύ ότι ο κύριος Πούτιν αποφάσισε να αποσύρει μεγάλο μέρος των στρατιωτικών μέσων που είχε εγκαταστήσει στη Συρία η Ρωσία. Επίσης, λάβαμε γνώση πρώτο βουλειών προερχομένων από ευρωπαϊκές χώρες που τείνουν ε, να φράξουν το δρόμο των Βαλκανίων για τους Σύρους πρόσφυγες και σαφώς επιδείνωση τις κατάστασης στην, ε, Ευρώπη, στην Ελλάδα μετά το κλείσιμο των συνόρων με την ε, Μακεδονία, λέει ο και ενδεχομένω και την Βουλγαρία. Επίσης, από πλευράς της Τουρκίας διατυπώθηκε αίτημα για την για τον διπλασιασμό των ποσών υποστήριξης που έχουν ενδεχομένως να ε, προσφέρουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων σε μια σύνοδο που πρόκειται να δεξαχθεί την επόμενη Παρασκευή ε, με την Τουρκία. Υπογραμμίζω και προσθέτω επίσης ότι παρά την πολιτική υποστήριξη και την οικονομική υποστήριξη που ε, υποσχόμαστε προς την Τουρκία, έχουμε ως Επιτροπή των Προϋπολογισμών τις επιφυλάξεις μας σε σχέση με την ε, με τις επιλογές Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλουμε ιδιαίτερως να υπογραμμίζουμε πως χρειάζεται να είναι πιο τακτικές οι επαφές. Η Επιτροπή μας ιδιαίτερως, αλλά γενικότερα το Κοινοβούλιο έχει την εντύπωση πως πολύ συχνά τις πληροφορίες συλλαμβάνει εκ των υστέρων. Αδυνατώντας έτσι να κάνει τίποτε περισσότερο από το να επικυρώσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου επί τη βάση βέβαια των προτάσεων της Επιτροπής. Επίσης, σε συνέχεια της αποστολής αυτής, μια νέα αντιπροσωπεία της Επιτροπής ε, των Προϋπολογισμών πρόκειται να μεταβεί στο Λίβανο και την Ιορδανία, σας είπα πότε ακριβώς, με τη δυνατότητα έτσι να, να συζητήσουμε τη συνέχεια που έχει δοθεί στις υποσχέσεις των ε, χορηγών, όπως αυτές εκφράστηκαν το Φεβρουάριο στο Λονδίνο και το ζήτημα αυτό των προσφύγων ασφαλώς θα αποτελέσει κύριο μέλημά μας και θα μας κινήσει στις εργασίες μας το υπόλοιπο του χρόνου. Ασφαλώς και στην α, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του πολιτισμού συνομικού πλαισίου. Τις πληροφορίες έχετε λάβει λοιπόν με την ε, γραπτή μας παρατήρηση. Έχετε ενημερωθεί λοιπόν. και υποχρεούμαστε να διατυπώσουμε κάποια, σαφ... κάποια σαφή μηνύματα. Γι' αυτό και με ευγνώμων προς τον Γκυγιόμ Ρέ, ο οποίος μαζί με την ομάδα του από τη Γραμματεία έκανε τη σχετική σύνταξη. Πρόκειται για μια έκθεση την οποία έχουμε ε, διαθέσει στα μέλη της Επιτροπής από την προηγούμενη εβδομάδα, ορισμένοι μεταξύ των οποίων ο Ερνέστ Μαργκάλο, ο Σκάιερ, έχουν διατυπώσει ήδη παρατηρήσεις και τις ενσωματώσαμε βέβαια στην έκθεσή μας. έτσι ώστε να ε, αποδοθεί μια αρκετά ε, ακριβή εικόνα των όσων είδαμε και επισκεφθήκαμε ένα καταβλισμό κοντά στο Καζιέντεπ όπου μας εντυπωσίασε η ποιότητα της ε, υποδοχής στον καταβλισμό αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι από τα 2,5 εκατομμύρια προσφύγων από τη Συρία, μόνο 250.000 έχουν ε, βρει κατάλημα σε αυτόν τον καταβλισμό και είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ε, ζουν ε, στα περίχωρα των πόλεων, κυρίως στις νότιας νοτιοανατολικές Τουρκίας, όπου, στις νότιες Τουρκίας, όπου υπάρχουν σοβαρά, σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα. Έως και 400.000 παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο υπό τις συνθήκες αυτές και η κατάσταση αυτή διαρκεί όταν υποδέχθηκε τους πρώτους πρόσφυγες η Τουρκία. Προβλεπόταν κατά πάσα πιθανότητα ότι θα ήταν στιγμιαίο το φαινόμενο και ότι ταχύτατα θα επέστρεφαν στις αιστείες τους οι πρόσφυγες αυτή από τη Συρία. Ωστόσο η κατάσταση ε, διαρκεί, επιδεινούμενη και έτσι το να μένουν παιδιά τέσσερα και πέντε χρόνια. Γιατί μπορεί να σκεφτόμαστε ότι... Γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε ότι εχθές εορτάστηκε ή τιμήθηκε καλύτερα η ε, πέμπτη επέτειος από τις πρώτες ε, ένοπλες συγκρούσεις το 2011 στη Συρία. Από αυτά τα, αυτούς τους κατοίκους λοιπόν της Συρίας 5-6 εκατομμύρια έχουν βγει από τη χώρα τους εντωμεταξύ. Βρίσκονται είτε στην Ευρώπη, είτε στην Τουρκία, τον Λίβανο, την Ιορδανία. Και αλλού, χωρίς να έχουμε πάντα ακριβείς πηγές. 4 εκατομμύρια υποστηρίζουν το καθεστώς του Μπασάρα Αλάσατ και 8 με 10 εκατομμύρια που μένουν μέσα στη Συρία είναι εκτοπισμένοι εσωτερικά και άρα είναι πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα. Με τις επιθέσεις στο Χαλέπι πριν από ένα μήνα, με τους βομβαρδισμούς, κάποιοι, ε, αρκετοί από αυτούς προσπάθησαν να φύγουν για να σωθούν στην Τουρκία, αλλά η Τουρκία τους έκλεισε τα σύνορα. Άρα πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε και για τον προπολογισμό την ανάγκη υποστήριξη με ε, βοήθεια των ε, εσωτερικά εκτοπιστέντων ε, σύρων μέσα στη Συρία. Και βέβαια πρέπει να μας απασχολήσει και το πότε μπορεί να ε, επανέλθει η ειρήνη στη Συρία. Αυτό πρώτα απ' όλα. Γιατί έτσι μπορούμε να αναιρέσουμε τους λόγους της μετανάστευσης και να αρχίσουμε την ανοικοδόμηση της Συρίας. Και εκεί θα πρέπει η Ευρώπη να αρχίσει να προετοιμάζεται και να κινητοποιεί τα απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη ανθρωπιστική και γεωπολιτική πρόκληση. Είχαμε πολλές επαφές με τις τοπικές αρχές. Ήμασταν για μια μέρα στην Άγκυρα και μια μέρα στο Γκαζιάντεπ. Όπου στην Άγκυρα συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης που έδειξαν μεγάλη αποφασιστικότητα και ανυπομονησία να εισπράξουν τις ε, τη βοήθεια που είχε εξαγγείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχές οι οποίες μάλιστα δεν παρέλειψαν να διατυπώσουν τις επικρίσεις τους για την βραδύτητα και την περιπλοκότητα των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απογοήτευσή τους πολλές φορές. Η Τουρκία βεβαίως ε, εισπράττει από την Ευρώπη 650 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο με το σύμφωνο το προενταξιακό, το προενταξιακό μέσο. Και πρέπει να διατυπώσουμε την παρατήρηση ότι κατά τα φαινόμενα τουλάχιστον η συγκυρία οικονομική είναι ευνοϊκή. Φτάνει κανείς ε, στην ε, Άγκυρα, βλέπει παντού ε, εργοτάξια, γερανούς κτλ. στην νότια Τουρκία για να πάμε στην Νότια Τουρκία πήραμε αυτοκινητοδρόμους τριών ε, λωρίδων κάθε φορά. Η ανάπτυξη υπολογίζεται στα 4%. Ε, βιομηχάνους έχει πολλούς η χώρα. Άρα παραξενευόμαστε που δεν μπορούν να, ελέγξουν, να δείξουν μεγαλύτερη επαγρύπνηση για να ελέγξουν την ε, μετανάστευση από τη δική τους ακτή προς την Ελλάδα οι Τούρκοι εν προκειμένου. Ακούσαμε λοιπόν ε, επικρίσεις. Εμείς σημειώσαμε ότι αν θέλει κανείς να προχωρήσει περισσότερο ταχύτερα χρειάζεται ε, εμπιστοσύνη και για να υπάρξει εμπιστοσύνη απαιτείται διαφάνεια. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με τον οποίο συναντηθήκαμε μας απάντησε ότι για να περάσουμε πιο γρήγορα μπορούμε απλώς και μόνο να αξιοποιήσουμε τις υπηρεσίες των ε, υπηρεσιο, των ε, οργανισμών όπως η BERT και η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, όπου εκεί απάντησα εγώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει και, 650 εκατομμύρια ευρώ κατά μέσον όρο, γιατί το 2015 ήταν ακόμα περισσότερα, αλλά υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία γκρόσο μόντο προσφέρει με τα δάνειά της περί τα 2 δις το χρόνο στην Τουρκία. Στην, ε, Τουρκία. Άρα έχουμε μια πραγματική εταιρική σχέση και ζητώ συγγνώμη που δεν ε, χαιρέτησα νωρίτερα την άφηξη της κυρίας Κάτι Πύρη, ηγήτρια της Τουρκίας για την Επιτροπή ΑΦΕΤ, η οποία είναι μαζί μας σήμερα. Και θα της δώσω βέβαια το λόγο σε ένα λεπτό. Προσπαθήσαμε να αντιληφθούμε λοιπόν το πώς θα προχωρήσει η οικονομική χρηματοδοτική διάσταση για Τουρκία. Οι εταίροι μας μας είπαν ε, ξεκάθαρα πως έχουν κάνει τις εκτιμήσεις τους και πως είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τις πιο κατεπίγουσες δράσεις. Συγκεκριμένα την ανέγερση σχολείων για να ε, προσφέρουν εκπαίδευση στις 400 με παιδιά που αυτή τη στιγμή δεν πάνε στο σχολείο. Επίσης, στον τομέα της υγειονομικής ε, φροντίδας. Υπήρχαν αισθήματα. Επίσης έχουν ε, υποχρεώσει καινούριο μάλλον, αρχίζουν να υποχρεώνουν τους Σύρους να εργάζονται, άρα θα μπορέσουν να συμμετέχουν πιο εύκολα στην οικονομική, στον οικονομικό βίο της χώρας. Εμείς έχουμε ζητήματα καταρχάς συντονισμού, πρέπει να ρυθμίσουμε. Πρέπει να πω ότι συναντηθήκαμε με όλους τους εκπροσώπους φορέων, καταρχάς των ε, αντιπροσωπιών και ε, πρεσβειών των κρατών μελών ε, που βρίσκονται στην Άγκυρα. Και είπαμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η μεγάλη πρόκληση είναι ο συντονισμός των δράσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των εθνικών αντίστοιχα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αποτελεσματικότητα θα σταματήσω προς το παρόν και θα παρακαλέσω την κυρία Πύρη αν ε, θέλει να λάβει το λόγο τώρα. Και μετά θα παρακαλέσω και τους αδέλφους που έλαβαν μέρος ε, στη συνεδρίαση να μας ενημερώσουν για τις δικές τους ε, εμπειρίες. Κυρία Πύρη έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και... Διάβασα την έκθεση με μεγάλο ενδιαφέρον Πιστεύω ότι έχει μηνύματα πολύ σημαντικά τα οποία θα πρέπει να τα μεταδώσουμε και πέρα από, την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Στέκομαι σε δύο από αυτά. Γιατί είναι ε, στόχοι τους οποίους θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Πρώτα απ' όλα, είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγεται και το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό, ότι δεν θα πρέπει να εστιάζουμε μόνο σε εκείνου που βρίσκονται στου καταβλισμού. Υπάρχουν εκατομμύρια Σύριοι οι οποίοι δεν βρίσκονται σε καταβλισμού στην Τουρκία και πώ μπορούμε να βοηθήσουμε τι κοινότητε που υποδέχονται αυτού του ανθρώπου. Είναι κάτι το οποίο διαπιστώσαμε επισκεπτόμενοι ε, πόλεις στην Τουρκία. Υπάρχουν πόλεις τις οποίες πάνω από το μισό του πληθυσμού είναι πρόσφυγες και πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή, αυτό το ευαίσθητο θέμα. Είναι ξεκάθαρο ότι κάτι πρέπει να γίνει εάν μιλάμε για ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων στο τοπικό πληθυσμό και αυτό θα είναι δύσκολο και επίσης ε, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα που δίνονται στην Τουρκία θα, δοθούν, θα αξιοποιηθούν ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο ε, βασικό μήνυμα στο οποίο στέκομαι είναι ότι αυτό το μέσο δεν μπορεί να, το χρηματοδοτικό δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό εάν δεν εμπλακεί και η, όχι μόνο η κυβέρνηση της Τουρκίας αλλά και η κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία. Είχαμε ε, αναδείξει την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη ρητορική και σε αυτό που ακούμε στην Βρυξέλλες, όπου ακούμε ότι τα χρήματα αυτά δεν πρέπει να φτάσουν στις ε, τουρκικές αρχές, πρέπει να ε, για να αξιοποιηθούν αποδοτικά, ενώ αν κανείς ακούσει τι λέγεται στην Τουρκία, οι ίδιες οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις λένε ότι ναι, αλλά για να αξιοποιηθούν αποδοτικά αυτά τα χρήματα θα ε, έπρεπε να μπορούμε να εμπλακούμε. Δεν λαμβάνω θέση ως το Προ το ποιο θα έπρεπε να είναι ο αποδέκτη των χρημάτων. Αλλά σε κάθε περίπτωση για να υπάρξει αποτέλεσμα πρέπει να συμμετέχουν ε, οι άνθρωποι, οι οργανώσει που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Έχουμε συζητήσει στην τελευταία ομέλεια το ζήτημα της Τουρκίας και γενικότερα το ζήτημα της προσφυγικής κρίσης πρόκειται να εξεταστεί η έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα προσπαθήσω να δω ε, εάν ε, μπορούμε να εισαγάγουμε κάποιες τροπολογίες προερχόμενες από την Επιτροπή Προϋπολογισμού σε αυτή την έκθεση για την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Με αυτά τα μηνύματα. Επίσης υπάρχει στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών μια ε, έκθεση που προετοιμάζεται για το ζήτημα της μετανάστευσης. Σε μεγάλο βαθμό αυτή η έκθεση αναφέρεται στην ε, Τουρκία και στο μέσο το χρηματοδοτικό. Θα πρέπει να φροντίσουμε να συντονιστούμε και με τους συναδελφούς εκεί, έτσι ώστε τα μηνύματά μας να περάσουν και στην έκθεση της έκθεσης της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών, η οποία θα ε, έρθει, θα ψηφιστεί περίπου την ίδια χρονική περίοδο. Επίσης, κάποια άλλα ερωτήματα προς την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Πώς σκοπεύετε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε ε, την κατάσταση μετά την αποστολή σας. Ε, λέγεται ότι το Συμβούλιο επιθυμεί ε, τα πρώτα τρία δισεκατομμύρια να εκταμιευτούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Συζητείται επίσης η ε, το ενδεχόμενο επιπλέον χρηματοδότησης. Ποιο θα είναι λοιπόν ο ρόλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, ποιο θα είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πώς θα ασκήσει τον ε, κοινοβουλευτικό τον έλεγχο του Κοινοβουλίου. Επίση. είναι ένα θέμα για το οποίο δεν βρήκα κάτι να αναφέρετε στην έκθεσή σας, αλλά εγώ όπως έχω καταλάβει, το ζήτημα του φίλου δεν έχει αντιμετωπιστεί και δεν υπάρχουν σχετικές προτάσεις από την Επιτροπή. Και όλο συζητάμε στο Κοινοβούλιο για την ένταξη της διάστασης του φύλου στους προϋπολογισμούς. Είναι ε, μάλλον ε, άστοχο το να μην υπάρχει καθόλου διάσταση του φύλου στην αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος. Σας ε, ευχαριστώ κυρία Πυρή και σας ευχαριστώ επίσης για τη συνεργασία που είχαμε με πριν ε, ξεκινήσει η αποστολή, πριν φύγουμε για την Τουρκία. Θα ήθελα να μοιραστώ με τους συναδέλφους κάτι που άκουσα από έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο που γνωρίζει καλά την κατάσταση στην Τουρκία. Μου είχε πει είναι ότι το πρόβλημά μας ότι δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο όραμα για το τι θα έπρεπε να γίνει. Και ως εκ τούτου δεν έχουμε κάποιες κατευθύνσεις, δεν γνωρίζουμε προς τα που πηγαίνουμε και επίσης συχνά υπάρχει και διγλωσία. Πριν ένα χρόνο επισκεπτόμενος στην Τουρκία διαπίστωσα ότι είναι δύσκολο να υλοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Οι διαδικασίες είναι περίπλοκες, χρειάζονται μήνες. Το Ταμείο Μαντάντ για τη Συρία δημιουργήθηκε αξιοποιώντας πόρους που είχαν περισσέψει από προηγούμενα ταμεία προενταξιακά ε, της περίοδου 2007-2013, αλλά ε, πολύ αργά ε, εκταμιεύονται αυτά τα χρήματα και αξιοποιούνται μόνο 40 εκατομμύρια μέχρι στιγμής. Επομένως, ενώ υπάρχουν ανάγκες επιτόπου, δεν καταφέρνουμε να δώσουμε τα χρήματα που χρειάζονται. Σας ευχαριστώ. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πιάνω τόπο τα χρήματα του προπολογισμού, έτσι. Επίσης είναι σημαντικό ότι έχουμε την κάτι εδώ και έτσι ακούμε τις ε, λεπτομέρειες του θέματος. Εγώ ήθελα όμως να σταθώ σε αυτό το τελευταίο που αναφέρατε όσον αφορά την υπόθεση των δύο φίλων θα πρέπει να διευκρινιστεί πως θα εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά που θα γίνουν με αυτά τα κονδύλια, η παρακολούθηση, έλεγε ότι όλα αυτά θα καλύψουν και γυναίκες και ανηλίκους πρόσφυγες και στην Τουρκία και αλλού. Αυτό σας τονίζω, να μην το ξεχάσουμε να μπορέσουμε αυτό να το εντάξουμε στο κείμενο. Κύριο Ντελάνο, νομίζω πρόεδρε ότι ήταν ε, εξαντλητική η ε, έκθεση των πεπραγμένων όπως κάνατε. Άρα θα πρέπει να δούμε όλη την ε, εικόνα. τρόπο συμβολική καλά πήγε η υπόθεση σε σχέση με το τι είδαμε, αλλά όμω αναδύονται πάρα πολλά άλλα ερωτήματα και αναρωτιέμαι σε σχέση με όλα αυτά που μας είπαν ε, οι τουρκικές ε, αρχές. Τι θα γίνει, τι, τι τροπή θα πάρουν τα, τα πράγματα σε σχέση με την τουρκική πολιτική. Γιατί είναι πάντα παρόν ο πρόεδρος. Έχει γίνει τώρα δικτάτορας. Που χαλιναγωγεί τα ΜΜΕ και δημιουργεί πολλά προβλήματα. Σωστά τα είπατε. Ότι πολλά πράγματα ε, γίνονται με τη λογική του βλέπουμε και κάνουμε. Όμως ε, εδώ μιλάμε για τον κοινωνικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό των κρατών μελών. Άρα πώς θα οργανωθούμε, ποιος τον αποδέκτης των κονδυλίων, με ποιο πρόγραμμα. Είναι πολλά τα ερωτήματα που τίθενται. Άρα το Κοινοβούλιο θα πρέπει να απαιτήσει να σχετιστεί με κάθε χρηματοδότηση για την ε, μεταναστευση και όχι μόνο για τα χρήματα του κοινωτικού προϋπολογισμού. Θα πρέπει επομένω να αναλάβουμε ρόλο συντονιστικό. Πριν προχωρήσουμε, από σήμερα κιόλας να κάτσουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Αυτό να το εγκρίνουν οι μη οργανώσεις και οι τουρκικές αρχές. Όντως ε, είναι αξιόλογα τόσα γίνονται εκεί. Αλλά θα πρέπει να κατευθυνθούν όπου πρέπει τα χρήματα, αλλά τα πράγματα να γίνουν οργανωμένα. Βάση προγράμματος, βάση πλάνου. Να δούμε πολλά κατά την αποστολή. Θα πρέπει επομένως να συνεχίσουμε στην ίδια ρότα. Εύχαστο λέει ο πρόεδρος και δίνει τον λόγο στον κύριο Φερνάντες. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για να λύσουν το πρόβλημα δεν αρκεί το να συστρατευτεί μόνο το σύνολο των κρατών Θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να ασχοληθεί. Βέβαια εμείς είμαστε ο πιο μεγάλος δωρητής και επίσης ε, εμεί είμαστε ε, αυτοί που θίγονται προς το αυτό το πρόβλημα, μια που εμείς υφίσταμε αυτή την εισαγωγικά εισβολή στα σύνορά μας, άρα θα πρέπει να συντονιστούμε, άρα θα πρέπει επίσης να αναβαθμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε. Θα πρέπει όμως να τηρούν και τα κρατημέλη τα συμπεφωνημένα. Αλλά πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλε συνθήκε για να προχωρήσουμε στην επίλυση του προβλήματο. Και το πρόβλημα είναι ότι τα κράτη-μέλη ακριβώ δεν τηρούν τα συμπεφωνημένα, άρα χρειάζεται ένα μηχανισμό να βοηθήσει του ε, πρόσφυγε ε, στην ε, Τουρκία. Είπαμε από τον κοινωνικό προπολογισμό θα διατεθούν τρία δι. Ένα δι από τα κράτη-μέλη και δύο από τον κοινωνικό προπολογισμό συγκεκριμένα. Αυτό όλο θα πρέπει να εκταμιευθούν. Και τα κοινωνικά δύο δι θα πρέπει να βρεθούν από άλλα κεφάλαια του υπροπολογισμού. Πολύ σημαντικό αυτό, γι' αυτό και το έχουμε επαναλάβει. Επανειλημμένα μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες. 10% είναι σε στρατόπεδα και 90% είναι εκτός αυτών των στρατοπέδων ή καταβλισμών. Είναι, ναι, μιλάμε για μια ολόκληρη χαμένη γενιά. Χρειάζονται παιδεία, χρειάζονται εκπαίδευση, κατάρτιση. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Δεν είναι δυνατόν να κατραγωθούν τα όνειρα μιας ολόκληρης γενιάς. Άρα θα πρέπει ο κοινωνικό προπολογισμό να χρησιμοποιηθεί και έτσι να εξασφαλίσουμε πως η γενιά τούτη ε, δεν θα χάσει το τρένο. Ή ακόμα χειρότερα δεν θα γίνει βορρά των εξτρεμιστών. Τώρα κάτι άλλο. Έχουμε πει πολλά για τους πρόσφυγες. Αλλά εν μέσω αυτών υπάρχουν και κάποιοι που δεν γίνεται να καταστούν πρόσφυγες και σας εξηγώ τι εννοώ. Πάρα πολλοί από αυτούς κάναν πρόθυμα τους πρόσφυγες γιατί αναζητούν την ασφάλεια. Πάρα πολλοί δεν μπορούσαν να ξεφύγουν, να βγουν από την Συρία και ακόμα είναι εκεί. Μιλούμε για 11 ε, εκατομμύρια Σύρων οι οποίοι συνεχώς ε, μετακινούνται, συνεχώς ε, μέρα και νύχτα εφίστανται επιθέσεις. Οπότε και εμείς εκεί επικεντρώνουμε τις προσπαθίες μας. Θα πρέπει να καλύψουμε αυτούς τους πρόσφυγες, αλλά να μην ξεχνούμε και το ότι χρειάζεται ένα ειρηνευτικό σχέδιο που να ωφελήσει εκείνους που δεν έχουν βγει από τη χώρα. Δηλαδή εκείνους που θα ήθελαν να είναι πρόσφυγες αλλά δεν τα κατάφεραν. Εγώ τους σκέφτομαι κάθε μέρα. Γιατί στα μάτια των προσφύγων είδα να αντικαθρεφτίζονται οι επιθυμίες αυτών που δεν μπόρεσαν να φύγουν, να ξεφύγουν. Άρα θα πρέπει να φροντίσουμε και αυτή τη γωνίτσα της ε, υδρογείου. Να βρούμε επομένως ένα ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο είναι αποτελεσματικό και γρήγορο. Επίσης, θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είπαμε ότι οι επενδύσεις, έχουμε ήδη επενδύσει δύο δις, θα πρέπει να γίνουν έργα υποδομής, σχολεία, για παράδειγμα τα οποία ακριβώς να φορούν τους πρόσφυγες. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια και οι περισσότεροι εξ αυτών δεν βρίσκονται στους καταβλισμούς. Άρα θα πρέπει να φροντίσουμε να γίνουν έργα υποδομής για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, θα πρέπει για όλα αυτά να υπάρξει σωστός συντονισμός και να μην ξεχνούμε τον ρόλο της Τράπεζας Επενδύσεων. Ευχαριστώ. Κύριε Μαραγκάλη, για το λόγο λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή η αποστολή πραγματικά βοήθησε για θετικά αποτελέσματα, ήταν χρήσιμη. Πραγματικά χρειάζεται. μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε τι γίνεται. Να έχουμε στοιχεία αξιόπιστα για το τι γίνεται εκεί. Και ακριβώς η έκθεση των πεπραγμένων είναι ακριβής, είναι πλήρης. Σίγουρα βέβαια είναι προσχετικές οι διατυπώσεις. Αναγκαστικά, καταλαβαίνουμε γιατί. Όμως, Θα πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι όπως το παίζουν και οι τουρκικές αρχές. Να ακούσουμε την επίσημη άποψη. Βέβαια πολλές φορές η επίσημη άποψη δεν αντικατοτρίζει πλήρως την αλήθεια. Δεν λέω ότι ψεύδονται, αλλά, αλλά πολλές φορές δεν αποτυπώνεται όλο το τοπίο σε αυτά που ακούμε. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται σαφώς ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται από οικονομικής πλευράς. Για τη σελίδα 4 αυτής της έκθεσης έχετε ένα πίνακα και εκεί βλέπουμε ότι αναφέρονται μέχρι 7 διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης. συμπληρωματικότητα, συντονισμός, αποτελεσματικότητα αυτών των πηγών χρηματοδότησης. Όλα αυτά θα πρέπει να δούμε πώς θα αποδώσουν. Άρα αυτό που χρειάζεται πρώτα πρώτα όπως είπαμε είναι όλα αυτά να τα σιγουρέψουμε ακριβώς σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης που αναφέρατε. Βλέποντας κάπως ευρύτερα τα πράγματα και στρατηγικά. Και να δούμε πρόθεσμα τι πρέπει να γίνει, τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, επίσης εδώ θα πρέπει να προσθεθεί κάτι. Τα κονδύλια από τα κράτη-μέλη. Ήρθαμε σε επαφή με τα κράτη-μέλη. Βέβαια ακόμα δεν γνωρίζουμε τι πόροι θα διατεθούν. Αυτά θα πρέπει να φροντίσουμε να πιστώσουμε εμείς. Να δούμε τι γίνεται με αυτό το 10% που βρίσκεται στους καταβλισμούς. Αξιολογούμε, θεωρήσαμε ότι είναι θετικός ο απολογισμός των όσων γίνονται. Ε, θεωρούμε ότι όλοι οι καταβλισμοί στο ίδιο επίπεδο. Αλλά τι γίνεται με το 90% εκτός καταβλισμών. Τεράστιο ερωτηματικό. Εκεί τι πληροφορίες να έχουμε. Καμία πληροφορία. Γνωρίζουμε ότι κάποιοι από αυτό το 90% Ε, είναι, ή τόσο κάποιοι από αυτούς, είναι αυτοί που φεύγουν Τουρκία για να περάσουν στην Ελλάδα. Δεν έχουμε όμως αξιόπιστες πληροφορίες για το τι κάνει η Τουρκία σχετικά με αυτό. Τι κάνουν, πώς φεύγουν από τη χώρα, από την Τουρκία. Τι ρόλο παίζουν οι μαφίες των διακινητών. Για να σα τα πω καλύτερα μισό λεφτάκι στα ισπανικά. Δεν ξέρω αν είδατε αυτές τις εικόνες τώρα, τώρα στο γιο αυτή τη βδομάδα, τι γίνεται στις τουρκικέ αρχές που είχαμε και ένα σκάφο με ανήλικους, με παιδιά και είχαμε επίσης την τουρκική εκτοφυλακή που χρησιμοποίησαν βία, σωματική βία κατά αυτών, αυτής της ομάδας. Τους βαρούσαν τους χτυπούσαν. Ε, αυτό είναι δείγμα της συμπεριφοράς των τουρκικών αρχών σε σχέση με τη διαδικασία της εξόδου των προσφύγων από την Τουρκία προς την Ελλάδα, ε, τότε νομίζω ότι βλέπουμε ένα κομμάτι της πραγματικής εικόνας που μας έλειπε. Τώρα, η τελευταία μου σκέψη, Πρόεδρε, να το πούμε ξεκάθαρα, κινδυνεύουμε ότι όταν καταφέρουμε να χωνέψουμε το τι γίνεται και το πόσα δαπανώνται, ποιος τα δαπανά, πού τα δαπανά, τότε να έχουμε μια κοινή στρατηγική, ένα πρόγραμμα δράσης ή κάτι τέτοιο, τότε θα μπορέσουμε να νοικοκυρέψουμε το τι κάνουμε, τις ευθύνες μας και τότε νομίζω ότι θα αλλάξουν τη ρότα των εξελίξεων, θα υπάρξει μια συμφωνία. Τότε θα μπορέσουμε να φρενάρουμε τις εξελίξεις, τη σύγκρουση, τον πόλεμο στη Συρία. ούτως ώστε αυτά τα 2,5 εκατομμύρια να έχουν ένα διαφορετικό αύριο ή τέλος πάντων να γυρίσουν στη χώρα. Όμως υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος για άλλη μια φορά να αργήσουμε και να μην δίνουμε την έγκαιρη σωστή απάντηση στο πρόβλημα. Γι' αυτό ήθελα να σας πω. Να σας επισημάνω το πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, αλλά όμως από την άλλη μεριά είναι εξαιρετικής ποιότητας ε, αυτό το οποίο ε, κάναμε στην Τουρκία, στην ε, Άγκυρα και στην Γκαζιαντέπ. Ο Πρόεδρος. Κύριε Μαργέλη, σε ευχαριστούμε. Κύριε Τζάνι, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρο που οι συναδέλφοι κλείνει το μικρόφωνο του μιλητή όμως. Μικρό, Συμφώνησαν με αυτή την πρότασή μας στους συντονιστές, την πρόταση που διατυπώσαμε από λίγους μήνες και έτσι αυτή η αποστολή απέδωσε χρήσιμα αποτελέσματα. Και εγώ συμφωνώ με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι, γιατί αυτή η εβδομάδα ήταν ε, πάρα πολύ εντατική και μπορέσαμε να έχουμε μια οπτική των πραγμάτων ευρύτερη για το τι γίνεται στην ε, Τουρκία και τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσουμε στην επίλυση αυτού του προβλήματος και να γίνει κατανοητό ότι αυτή η συνεννόηση κρατών μελών και Τουρκίας σήμερα ε, είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Τα εξήγησε πάρα πολύ καλά ο συνάδελφος Μαραγκάλη. Μας δίνεται η εντύπωση του πώς μας τα λένε οι τουρκικές αρχές και έχουμε αυτά τα τρία πόσο είναι, 6 δις, όσα και αυτά που θα δώσουμε, θα πρέπει να αποκτήσουμε τη βεβαιότητα για το πώς θα διατεθούν αυτά τα χρήματα. Στις επαφές μας με τις τουρκικές ε, αρχές, ε, στις διαπιστώσεις που κάναμε, δεν πρόκειψε η βεβαιότητα για το πώς θα διατεθούν αυτά τα χρήματα. Και είδαμε ότι πολλές φορές ε, αλλιώς μας τα έλεγαν. Και το μήνυμα πολλές φορές ήταν δώστε μας τα λεφτά και εμείς σας πολύ νοιάζει για το πώς εμείς θα τα αξιοποιήσουμε. Κρίμα μόνος που κατά αυτές τις διαπραγματεύσεις η αρμοδιότητα της Επιτροπής μας δεν μπορούσε να είναι τέτοια που να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. γιατί ακριβώς διαπιστώσαμε το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι επαφές και διαπραγματεύσεις. Πριν από την αποστολή δεν είμαι καθόλου σίγουρος για το κατά πόσον το πιο σημαντικό στην υπόθεση αυτή είναι τα χρήματα. Δηλαδή για να διαχειριστούμε καλύτερα τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μετά ε, την αποστολή είμαι ακόμα λιγότερο σίγουρος για το τι θα γίνει και πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Έχουμε άλλωστε και αυτή την έκθεση του 2009 του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τους πόρους που διαθέσαμε τότε. Γι' αυτό σας λέω, δεν βλέπω να έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό, αλλά μακάρι τα κράτη-μέλη να κάτσουν για να σκεφτούν καλύτερα το πώ θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα, είτε είναι 3 είτε είναι 6 δι. Και να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίξει πιο σημαντικό ρόλο και εμεί εδώ στην Επιτροπή μα όσον αφορά το πώ θα διαμορφωθεί η κατάσταση για την αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων. Από ό,τι είδα πάντως μάλλον Καλύτερα να δώσουμε αυτά τα χρήματα στην ε, Ελλάδα που έχει τόσο μεγάλα προβλήματα με τις ε, μεταστατικές ροές και έχει και τόσο μεγάλα δημιουργικά προβλήματα όπως είναι γνωστό. Ίσως θα δώσουμε στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία. Και έτσι ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερο έλεγχο ως ευρωπαϊκές αρχές επί της αξιοποίησης αυτών των κονδυλίων. Α κάτσουμε και να σκεφτούμε πώς θα επενδύσουμε αυτά τα χρήματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι εκτό αυτή. Αυτά είδαμε εκεί στους ε, καταβλισμούς. Και επίσης τι έγινε το καλοκαίρι στις ακτές της Σικελίας δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πώς έχουν τα πράγματα. Δεν μπορεί κανείς να ανασχέσει αυτές τις μεταστητικές ζωές. Τι να κάνει στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για το... Αν μπορεί κανείς να σταματήσει το, το νερό. Μα το νερό, μου το βάλουμε ένα εμπόδιο, θα το παρακάμψει γύρω-γύρω. Μιλάμε για άτομα τα οποία θέλουν να γλιτώσουν από πόλεμο, από ακραία φτώχεια, οπότε οποιαδήποτε σκέψη κλεισίματος ε, ε, συνόρων δεν θα ωφελήσει και θα συνεχίσουν αυτοί οι άνθρωποι να ψάχνουν τη σωτηρία. Κάπου, κάπου να αναζητούν ένα γυροβόλιο σε κάποια πιο σίγουρη χώρα. Οπότε γι' αυτό σας λέω, η μόνη λύση είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες ε, ειρήνης, ανάπτυξης, αρμονίας στις χώρες εκείνες. Αυτό μας λέγανε τους ε, καταβλισμούς. Πέστε μας πώς θα γυρίσουμε στα σπίτια μας. Αυτό προσδοκούν. Άρα, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί εκεί και όχι στην Τουρκία. Εκεί να δούμε τι επενδύσεις και τι αναπτυξιακές ενέργειες μπορεί να γίνουν τόσο να τους δώσουμε την ευκαιρία σε εκείνους να γυρίσουν στη χώρα προέλευσης. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Καγιά. Ευχαριστώ. Δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος όσο οι συνάδελφοι που έλαβαν το λόγο. Γιατί δεν είναι ούτε συμφωνημένο ούτε και στόχος των ε, ποσών αυτών να υποστηρίξουν το τουρκικό κράτος. Ας κοιτάξουμε από ποιες γραμμές του προϋπολογισμού προκύπτουν τα ποσά αυτά. Η δική μας συμβολή δηλαδή στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για το ε, ΙΠΑ είναι κομμάτι για την ανθρωπιστική βοήθεια και τίποτε δεν μας εμποδίζει να διαθέσουμε τα κονδύλια αυτά στις ίδιες τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες βρίσκονται στους καταβλισμούς και δουλεύουν με τους πρόσφυγες. Βεβαίως θέλω και πιστεύω ότι θα έπρεπε ε, να δώσει το σώμα μεγάλη σημασία και έμφαση στο θέμα αυτό, να πάει στο παγκόσμιο πρόγραμμα, ε, το επιστηστικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών το ποσό που θα εγκρίνουμε και να διατεθεί απευθείας στους καταβλισμούς με βέβαια χαμηλότερο και κόστος ε, διαχειριστικό. Είδαμε ότι υπάρχουν 300 περίπου εργαζόμενοι στο Οσμάνιε για να στηρίξουν το παγκόσμιο πρόγραμμα. Άρα λοιπόν παγκόσμιο, πρόγραμμα, ε, παγκόσμιο επιστητικό ε, UNICEF για τα σχολεία. Ε, πράσινη, Ερυθράη, Μισέλινος. Όλες αυτές οι οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται και βοηθούν τους πρόσφυγες χωρίς να χρειάζεται να παρεμβαίνει η τουρκική κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να δώσουμε καμία λευκό επιταγή στον Ερντογάν. Και το ζήτημα και μόνο της διοχέτευσης των κονδυλίων στην Τουρκία μπορεί να αποτελέσει για μας μια εγγύηση για το πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Με την αντιπροσωπεία, εγώ αντιλαμβάνομαι πως η ΑΦΑΤ, ΑΦΕΤ η Υπηρεσία για την Αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών της Τουρκίας παρακολουθεί ιδιαίτερα την ε, κατάσταση. Είναι ωστόσο μια υπηρεσία η οποία υπάγεται στην προεδρία της δημοκρατίας. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε με πολύ μεγάλη προσοχή αυτή η ΑΦΕΤ, η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών ε, και λοιπόν να ε, ελέγχεται ως προς την διαχείριση των κονδυλίων. Και όπως είπε και η Κάτι Πύρη, τα κονδύλια για την υποστήριξη των προσφύγων πρέπει να δίνουν και έμφαση στην κατάσταση των γυναικών σε έναν βαθμό νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταφέρει. Δεν λέω ότι δεν ε, μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά εάν δούμε πόσο ιστερικές ε, συζητήσεις γίνονται στην ε, Γερμανία για το κατά πόσο θα πρέπει τα χρήματα να φτάνουν ως, ως χρηματικό ποσό ή εάν θα πρέπει να προσφέρονται ως υπηρεσία και το γεγονός ότι η ΑΦΕΤ μπορεί να διαθέτει κορδίλε με τη μορφή μιας κάρτας στην οποία αποφασίζει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος πρόσφυγας πώς θα διαθέσει να αγοράσει φερρυπίν, χρήμα, ε, να αγοράσει τρόφιμα μια γυναίκα για την οικογένειά της είναι μια κατεύθυνση στην οποία μπορούμε παραπάνω να εργαστούμε. Και τελευταία παρατήρηση και παρακαλώ την Επιτροπή να μας υποστηρίξει αυτό, με ιδιαίτερα, με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα τα μεγέθη στις ε, περιοχές της παραμεθόρες ιδιαίτερως αναλογίες προσφύγων σε σχέση με κατοίκους στην Βόρεια Βεσφαλία, Ρινανία, από την οποία προέρχομαι εγώ, ο λόγος είναι 80 προς 1. 80 κάτοικοι για ένα πρόσφυγα. Στην ε, Τουρκία είδαμε λόγο μέχρι και 1 προς 1 ή 11 προς 10. 11 πρόσφυγες για 10 Τούρκους υπαλλήλ, ε, υπηκόους, συγγνώμη. Μην ξεχνάτε και όλες τις λοιπές υπηρεσίες που συνεπάγεται αυτό. Είτε πρόκειται για αποκομιδή σκουπιδιών, είτε πρόκειται για σχολεία, είτε πρόκειται για διατροφή. Όλα αυτά τα πράγματα και βέβαια λαμβάνουμε υπόψη τα κονδύλια της προενταξιακής βοήθειας ε, που πάνε στην Τουρκία για να υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτή, αλλά πρέπει οπωσδήποτε τα χρήματα που θα διατεθούν να πάνε στους πρόσφυγες για να τους υποστηρίξουν. Δεν ξέρω εάν πάνε στην κεντρική κυβέρνηση, εάν, πάνε στις, ε, αν πρέπει να πάνε στις ε, τοπικές αρχές, επαρχίες, ε, νομαρχίες κτλ. Ή αν μπορούμε πολύ πιο συγκεκριμένα να στοχεύσουμε τις εμπλεκόμενες τοπικές κοινότητες για να διατεθούν εκεί κατευθείαν τα χρήματα. Πάντως θα παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα να μεριμνήσει για τον στόχο αυτόν. Και αγαπητοί συνάδελφοι, ένα πράγμα ας, πρέ, σταματήσουμε, μην γυρνάμε ο καθένας στη χώρα μας λέγοντας «Α, τα χρήματα αυτά τα σπαταλάμε, αυτά τα χρήματα είναι μια λευκό επιταγή για τον Ερτογάν. Α σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό. Είναι χρήματα για να φροντίσουμε του πρόσφυγε και το ταχύτερο δυνατό, αλλά και το πλέον άμεσο δυνατό πρέπει να φτάσουν στου ανθρώπου αυτού. Να κάνουμε και εμεί σωστά τη δουλειά μα. Ευχαριστώ. Έχω δύο ακόμα συναδελφούς που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα σας ζητήσω να μην μακρογορήσετε γιατί έχουμε πολλούς. Θα προσπαθήσω, λέει η κυρία Νεριάντα, να είμαι σύντομη. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του συναδέλφου Γιούνης γιατί δεν μπορούσε να είναι παρόν σήμερα παρά το γεγονό ότι συμμετείχε στην αποστολή. Είναι ασθενής. Ε, ε, υποστηρίζει όμως την έκθεση. Συμφωνώ με τον κύριο Μαραγκάλ και άλλους συναδέλφους, πρέπει να έχουμε μια πρακτική, πραγματιστική προσέγγιση και να δούμε πώς αυτά τα χρήματα θα βοηθήσουν για την εκπαίδευση, για την ασφάλεια, ιδίω των γυναικών και των παιδιών. Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά και οι γυναίκες είναι από πρώτα θύματα και ιδιαίτερα ευάλωτοι ε, ομάδες προσφύγων, ιδιαίτερα κινδυνεύουν από σεξουαλική βία και επίσης χρειάζεται να καταλήξουμε σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο ουσιαστικό. Γιατί διαφορετικά δεν αντιμετωπίζουμε την ε, αιτία ε, που δημιουργεί αυτού του πρόσφυγε τη γενεσιουργό αιτία. Πρέπει να επιληθεί στη σύγκρουση ε, στη Συρία Πρέπει ταυτόχρονα να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις πολιτικές του καθεστώτος Ερτογάν, τι επιθέσεις κατά των Τούρκων, τις επιθέσεις κατά της ελευθερίας του τύπου. Επομένως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και αυστηροί έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα κονδύλια που δίνουμε σωστά και για το λόγο που τα δώσαμε και οφείλουμε και ως Επιτροπή Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι ε, εντάσσεται στις αρμοδιότητές μας για να ε, βεβαιωθούμε ότι τα κονίλια χρησιμοποιούνται όπως πρέπει. Ευχαριστούμε. Γέτεμακη. Κυρία Γέτεμα. Η κυρία hyvin tehdystä raportista. Tämä Ευχαριστώ πολύ. Σας συγχαίρω για αυτή την εξαιρετική έκθεση που δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται κανείς. Ο στόχος της αποστολής ήταν να δούμε τι είδου και πόσοι πόροι χρειάζονται. Και πιστεύω ότι μετά από αυτή την αποστολή έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Γι' αυτό ήταν κατά την άποψή μου ορθό να στείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια τέτοια αποστολή για να δει η διεισόμαση πως χρησιμοποιούνται τα χρήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεισφέρει έτσι στον διάλογο στη συζήτηση που γίνεται. ακούγεται ή λέγεται μερικές φορές ότι τα χρήματα τα δίνουμε στην Τουρκία ή τα χρήματα τα δίνουμε στον Ερντογάν. Όχι. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτά τα χρήματα δίνονται για ανθρωπιστική βοήθεια. Ότι τα χρήματα αυτά τα δίνουμε για ε, να βοηθήσουμε ανθρώπους και αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για το πώς ε, χρησιμοποιούνται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι χρήματα για την Τουρκία ή για τον Ερντογάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη στο σπορ του να ξοδεύει χρήματα χωρίς διαφάνεια. Επομένως, πώς κουνάμε εμείς το δάχτυλο στον Ερτογάν. Νομίζω το επόμενο βήμα που πρέπει να ακολουθήσει μετά από αυτή την αποστολή είναι το εξής. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία θα πρέπει να τις δοθεί η δυνατότητα ε, και να τους δοθούν οι απαραίτητοι πόροι για να το πράξει αυτό, να αξιολογεί ε, και να παρακολουθεί την κατάσταση με τους πρόσφυγες. Είναι δυνατόν η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία να μην γνωρίζει ποια είναι η πραγματική κατάσταση, να εκπλήσεται που υπάρχουν προσφυγικοί καταφλισμοί, να μην αντιλαμβάνεται την ανάγκη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι άνθρωποι που βρίσκονται επί τόπου πρέπει να έχουν πολύ καλύτερη εικόνα. Αυτό που χρειάζεται είναι επιστημιστική βοήθεια και εκπαίδευση. Η UNICEF έχει τεράστια εμπειρία στο να παρέχει τέτοιου είδους ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η αποστολή και νομίζω ότι η έκθεση καταγράφει πιστά τα ευρήματά μας, τις διαπιστώσεις μας, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει και να εκφράσουμε τις εντυπώσεις μας με τρόπο εύκολο και μπορούμε ίσως να πλησιάσουμε και τις κυβερνήσεις μας με τον τρόπο αυτό γιατί πολλές φορές διερωτώμεθα τι είδους προτεραιότητες ε, τους ε, κινούν, τις κινούν, πώς δεν βλέπουν την πραγματικότητα όταν έδωσαν τόση σημασία για τον Brexit και ανέβαλαν ε, συζητήσεις και αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το προσφυγικό και την Τουρκία. Όσο σημαντικό και είναι το Brexit. Για την κυρία ε, Πύρη και τις ε, ερωτήσεις. Βεβαίως έχουμε αρμοδιότητες κοινοβουλευτικές που σκοπεύουμε να ασκήσουμε. Η διάθεση του μηχανισμού για την διάθεση και τα εμβάσματα τα οικονομικά, τρία δις, έξι δις δεν ξέρουμε ακόμα, εμείς θα μεριμνήσουμε να ασκήσουμε τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές μας για να παρακολουθήσουμε πώς θα προχωρήσουν τα χρήματα αυτά και αντλούμε και τα σχετικά διδάγματα και εν ώψη της αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, τη μεσοπρόθεσμη γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα δημοσιονομικό το οποίο έχει σχεδιαστεί για την ε, μπουνάτσα, για τα ήρεμα νερά και χρειάστηκε να αυξηθούν τα κονδύλια του τμήματος 4-3 ποιο ήταν κατά 25% από τον αρμόδιο συγγητή όταν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε κατεπίγουσες κρίσεις. Γι' αυτό λοιπόν σας διαβεβαιώ κυρία μου πως θα μεριμνήσουμε και θα επαγρυπνούμε πάντοτε στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και των δικαιωμάτων μας. Και προβλέπουμε ακόμα μια αποστολή στην Ιορδανία και τον Λίβανο. Τον Ιούλιο σκοπεύουμε να επισκεφθούμε την Ελλάδα για να δούμε και εκεί η μας την κατάσταση. Έτσι λοιπόν εάν έχει αναγερθεί τείχος ε, μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει με τη Λαμπεντούσα και την Σικελία. Και ευχαριστώ τον κύριο Τζίλη για την ε, πρόταση για την επίσκεψη στην Ιταλία και βέβαια και την ε, Τουρκία φέτος για τις γυναίκες. Στην επίσκεψή μας στο Κασιαντέπ θελήσαμε να επισκεφθούμε ένα σχολείο στα περίχωρα του Καζιαντέπ και όχι μέσα στον ε, καταβλισμό που μας δείξανε. Στο σχολείο λοιπόν αυτό είδαμε να διδάσκουν γυναίκες. Ασφαλώς μεταξύ των σύρων προσφύγων είναι πολύ, πολλές οι γυναίκες δασκάλες καθηγήτριες. Είδαμε λοιπόν να διδάσκουν ε, γυναίκες στο σχολείο αυτό που είχε ανεγείρει η ε, UNICEF. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι ιδιαίτερα μεριμνούμε για την θέση των γυναικών και σε αυτές τις δράσεις που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητήσαμε επίσης πίνακα των ενισχύσεων από Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη-μέλη, γιατί δεν έχουμε μια συνολική εικόνα του τι πράττουν και τι μπορούν να πράξουν η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα κράτη-μέλη στο τομέα αυτών. περιπτώσει, σταματώ εδώ. Την έκθεση μας θα τη διαβιβάσουμε στον πρόεδρο Σούλτς και ελπίζω οι αρχές μας, είτε, είτε κυβερνητικές είτε ευρωπαϊκές, να λάβουν υπόψη αυτή την έκθεση, που πάντως αποτελεί ένα για ιδιαίτερη επαγρύπνηση. Κυρία Καβίνιο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας κάποια σχόλια που εγείρονται από τη συζήτηση που έλαβε χώρα τώρα. Και γυρνάω στα αγγλικά. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τις ολόθερμες ευχαριστίες μου και να καλωσορίσω την ε, συζήτηση που έλαβε χώρα για την ε, ε, Επιτροπή, για την αποστολή της, για την έκθεση. Ιδιαίτερα θερμά ευχαριστούμε. Είναι πολύ ευπρόσδεκτη η συζήτηση λοιπόν που έλαβε χώρα γιατί δείχνει στεναρή, ομόφωνη θα έλεγα, υποστήριξη της Επιτροπής σας για έναν προφανή και ε, στεναρό ρόλο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κρίσης η Επιτροπή. Η αποστολή αυτή πιστεύω σας επιτρέπει σε εσά προσωπικά, αλλά θα μεταφερθούν τα ευρήματά σας, να αντιληφθείτε ποια είναι η κατάσταση στην Τουρκία και βέβαια σύμφωνα με τις προσεγγίσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπής, όπως απεδείχθη τι τελευταίες εβδομάδε και μήνε, ε, ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπιση. Και έτσι, σαν πρώτο σχόλιο, ευχαριστώ πολύ και εκφράζω την υποστήριξή μου στην προσέγγιση της Επιτροπής. Δεύτερον, Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να διαρευνά κάθε δυνατή πηγή και ευελιξία στα όρια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και του δημοσιονομικού καρονισμού. Αργότερα σήμερα θα κληθούμε να συζητήσουμε άλλες δράσεις στον ανθρωπιστικό τομέα. Αλλά η προσέγγιση μας είναι σαφέστατη. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε περιθώριο ευελιξίας. πιστεύματα και είπα προενταξιακό μέσο για την Τουρκία είναι δύο από αυτούς τους πόλους ε, ευελιξίας γιατί επιτρέπουν τη συλλογή κονδυλίων ευρωπαϊκών. Ο κύριος Μαραγάλ νομίζω ήταν εκείνος ο οποίος είπε πρέπει να αποφύγουμε επικαλύψεις και επαναλήψεις των ίδιων παρεμβάσεων ή απουσία συντονισμού. Αντιθέτως λοιπόν με, τα και, με το καταπίστευμα και το προενταξιακό μέσο μπορούμε να ε, συλλέξουμε σε έναν χώρο τα κονδύλια και να παρακολουθήσουμε την διαθεσή τους. Επίσης μπορούμε να εξασφαλίσουμε και προσέλκυση ε, χορηγιών και από άλλους χορηγούς. Για δεν το είπα, σημειώνω ότι υπάρχει δέσμευση και υποχρέωση των κρατών μελών να συμβάλλουν και εκείνα στην κατεύθυνση αυτή. Άρα και ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός και άλλοι χορηγοί ε, διαθέτουν τα κονδυλιά τους στο ίδιο ταμείο και επίσης βέβαια επιτρέπεται έτσι ο συντονισμό των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών στην χώρα και εδώ σημειώνω ιδιαίτερα το δικό σας ε, αίτημα να, έχει, να έχουμε μια πλήρη εικόνα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι κάνουν τα κράτη-μέλη ε, έχουμε προχωρήσει σε αυτό. Ακόμα δουλειά μένει να γίνει ασφαλώς, αλλά νομίζω ότι ε, είμαστε στο δρόμο. Η τρίτη μου παρατήρηση σχετική με κάποια από τα σχόλια που έγιναν σχέση με την αλλαγή συνθήκων και όντως αυτά που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες είναι ότι εξελίσσονται οι προκλήσεις, αλλάζουν μέρα με τη μέρα οι συνθήκες και προσπαθούμε να επιλύσουμε προβλήματα σε ένα σημείο για να διαπιστώσουμε ότι εμφανίζονται άλλα σοβαρά σε κάποιο άλλο. Άρα χρειάζεται ταχύτατη δράση. Ξέρω ότι έχει κάποιε επιφυλάξει σχέση με ορισμένα μέσα από αυτά που αξιοποιούνται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά η ανάγκη για ταχύτατη δράση νομίζω να γνωρίζεται ομόφωνα. Όπω η χρήση μέσων, αντί, ε, Φερρυπίν ε, το είπα, το πρωταξιακό μέσο για την Τουρκία, είναι σημαντικά μέσα για να συμπληρώσουν οποιασδήποτε άλλες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρισκόμαστε τώρα σε μια εβδομάδα που πρόκειται να γίνει και η Σύνοδος Κορυφής, άρα θα ληφθούν τις αποφάσεις συμπληρωματικές των όσων είπαμε σήμερα, αλλά εμείς θα τηρούμε πάντοτε πλήρως ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε εξέλιξη. Τελευταία παρατήρηση για την ε, ε, υλοποίηση στη χώρα την ίδια και με ενδιαφέρον παρακολούθησα σχόλια που ακούστηκαν σήμερα σε σχέση με την ανάγκη να εστιάζουμε στην, ε, ε, στον στόχο της διάθεσης των κονδυλίων ακριβώς εκεί που χρειάζονται, να γίνεται η διαχείρισή του σωστά, να γίνεται ακριβώς εκεί που είναι ανάγκη και για τον στόχο για τον οποίο έχουν προβλεφθεί. Σε αυτό δίνετε μεγάλη έμφαση και εσείς και βεβαίως θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε πως ε, το μέσον αυτό δεν είναι χρήματα για την Τουρκία. Το υπεγράμμισαν ορισμένοι εξημών, το υπογραμμίζω και εγώ για άλλη μια φορά. Δεν πρόκειται για μεταφορές κονδυλίων προς την τουρκική κυβέρνηση. Πρόκειται για χρήματα που στόχο έχουν να χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένες δράσεις στη χώρα και άρα υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για το, να, ε, για, για το πώς θα ληφθούν οι αποφάσεις πού θα διατεθούν τα κονδύλια αυτά. Βεβαίω και το Κοινοβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τα έργα αυτά, για την υλοποίηση, για το προϊόν που προκύπτει. Υπάρχει βεβαίω ήδη διαδικασία ενημέρωση, αλλά και εμεί διαρκώ σα προβα... υποβάλλουμε τι προτάσει και τι εξηγήσει. Ασφαλώ και δεν πρόκειται για, ελευ... για ελευκό επιταγή. Συμφωνώ απολύτω με όσα είπε ο κύριο Γκάιερ. Καθήκον δικό μα τη Επιτροπή αλλά και του Κοινοβουλίου <laughs> είναι να μεριμνήσουν όντως να μην είναι μία εν λευκό επιταγή και να υλοποιούνται τα σχέδια όπως ακριβώς έχουν προβλεφθεί. Με τα κονδύλια που έχουν προβλεφθεί και εκεί που έχουν προβλεφθεί. Και αν μου επιτρέπετε θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκίνεφ, συνάδελφα από την DG Near, ε, αρμόδια για το μέσον για την ε, Τουρκία για να σε εξηγήσει πολύ, πιο συγκεκριμένα την κατάσταση. Ο πρόεδρος, δεν θα είναι πάλι με την κυρία Τζόρτζεβα, δεν θα υπάρχει πάλι. Αυτό με ρωτάτε αν θα έρθει η κυρία Τζότζεβα. Μα δεν θα είναι αυτό και στο επίκεντρο των συζητήσεων με την κυρία Τζότζεβα. Όχι, όχι, διότι η ενημέρωση έχει να κάνει με ανθρωπιστική βοήθεια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το Turkish Facility, το μέσον για Τουρκία, έχει να κάνει με τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Τουρκία. Καλώς μια σύντομη ενημέρωση, παρακαλώ. 17 Φεβρουαρίου έγινε η πρώτη συνάντηση των κρατών μελών ε, για το μέσο για την Τουρκία και κατά τη συνάντηση εκείνη ζήτησαν τα κρατημέρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήταν στη συνάντηση να επιταχύνει του ρυθμού τη ε, υλοποίησης αυτής της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 την συμμετοχή για το μέσο. Στι 4 Δευτέρου υπεγράφησαν δύο συμβάσει μια για πιστική βοήθεια προς τους ε, πρόσφυγες και υπήρχε και μια σύμβαση με την UNICEF ούτως ώστε να καλυφθούν 100.000 ε, ανήλικοι όσον αφορά την φοιτησή του στο σχολείο. Τώρα, όσον αφορά τη διάσταση των δύο φίλων, την ισότητα των δύο φίλων, θέλω να σας πείσω την προσοχή στο άρθρο 3, παράγραφος 4 της σχετικής απόφασης μας εκεί, ορίζεται ξεκάθαρα ότι η διάσταση του φύλου όχι μόνο θα ληφθεί υπόψη, αλλά και θα προβληθεί σε κάθε φάση εφαρμογής του μέσου για την Τουρκία. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε και την κυρία Καλβίνιο για την ενημέρωση. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολύ στενή θα είναι η συνεργασία μας. για πρόσφυγες, έλεγχο των ε, μεταναστών και ευελπιστώ να επιστρέψει η, η ειρήνη στις περιοχές εκείνες γιατί αυτή είναι η ρίζα του προβλήματος. Τώρα βέβαια είμαστε 40 λεπτά πίσω από το χρονικό μας πλαίσιο και να δώσουμε τώρα το λόγο στη κυρία Καρδία Θάμπαλ για αυτό το κατάστημα για την Αφρική για να καλύψουν το χαμένο έδαφος πρόεδρε γιατί όπως ξέρετε τα πράγματα εδώ είναι πάρα πολύ σφιχτά ε, όσον αφορά την γνωμοδότησή μας, στην οποία προσπάθησα να ενσωματώσω τέσσερις βασικές αρχές. Πρώτα-πρώτα θέλουμε να υπάρχουν κάποιο είδους ε, μέσα, εργαλεία για να μπορούμε να ελοποιήσουμε αυτά τα οποία θέλουμε. Καταρχήν ήταν λοιπόν θετική η απόφαση, αλλά υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση αυτών των καταπιστευμάτων. Οπότε η σχετική πόρη δεν είναι δυνατόν να κατευθυνθούν προς άλλες πολιτικές, άλλες σε σχέση με το τι έχει προβλεφθεί στην αρχή. Άρα χρειάζεται στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής των κονδυλίων διαφάνεια και αυτό και κάνουμε. Οπότε θα πρέπει τα κρατή μέλη να εισφέρουν σε αυτό το καταπίστευμα αυτό που τους αναλογεί. Και αν δεν κάνω λάθος, είχαμε 81 εκτός από τα αρχικά 800 εκατομμύρια. Γενικώ πώς θα πρέπει να κάνουμε κάποια αξιολόγηση όπως προέκυψε και στην προηγούμενη συζήτηση γιατί έχουμε τώρα κάποια νέα μέσα, νέα εργαλεία τα οποία ad hoc επινοούμε. Φαίνεται επομένως ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι ούτε αρκετά ευέλικτο, ούτε προβλέπει αρκετά κονδύλια. Να, το συμπέρασμα της γνωμοδότησης. Άρα χρειάζεται για άλλη μια φορά μια αναθεώρηση του χρηματοδοτικού πλαισίου. Να, οι περιπτώσεις που αποδεικνύουν ότι χρειάζεται μια τέτοια αναθεώρηση. Γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες, ενώ το δημοσιονομικό πλαίσιο στενό εν κατακλείδη σαν παρατήρηση. Όλα αυτά τα ad hoc μέσα και εργαλεία τα προωθούμε ε, από πλευράς μας και θα πρέπει να προσέξουμε να μην απονευρώνουν ρόλο και τι αρμοδιότητέ μα ω Επιτροπή. Σα ευχαριστούμε που ήσασταν τόσο σύντομοι, λέει ο Πρόεδρο. Ποιο θέλει τώρα, ο κύριο Μπέγκε. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υποστηρίξω οπωσδήποτε και ρητά το βασικό μήνυμα ότι θέλουμε να τηρείται ο προπολογισμό όπως προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας και να εκτελείται έτσι. Υπάρχουν πολλές πολυάριθμες επιθέσεις και απόπειρες να αλλάξει αυτό, καθώς υπάρχει προσπάθεια να περιοριστούν, να περισταλούν οι αρμοδιότητες οι δημοσιονομικές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το άρθρο 122 παράγραφος 2 που έχει να κάνει, ε, βλέπουμε να ε, προσβάλλεται με τη δημιουργία του μηχανισμού ε, σταθεροποίησης, μετά στο 122.1 τώρα λένε θα ενημερώνεται το κοινοβούλιο. Και εδώ έχουμε να κάνουμε όχι μόνο με διαχείριση κονδυλίων, αλλά ακόμα και με επιλογές εξωτερικής ανάθεσης ε, υπηρεσιών που προσφέρεται στο ίδιο το κοινοβούλιο. Όταν λοιπόν η καιρή είναι δύσκολη, πρέπει κανείς πιστεύω να είναι σε θέση να ε, προσφέγει προσφεύγει στην χρήση κονδυλίων και εκτάκτων. Βεβαίως εν προκειμένου, αν θέλουμε να αναβάλουμε ή να αποφύγουμε την αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού σχεδίου, βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι παραγωνίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά τότε τι θα γίνει σε σχέση με την παγίωση μιας της πολιτικής, οπότε τα κράτη-μέλη θα δίνουν όλο και λιγότερα ή ελάχιστο ποσό στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και θα λένε άρα εμείς μπορούμε στη συνέχεια όποτε χρειαστεί να ελέγχουμε το πού θα πάνε τα λεφτά. Γιατί θα χρειάζεται πάντα να συμπληρώνεται ο προπολογισμό. Ε, είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παραμείνει ε, διατεθειμένο να εγκρίνει ένα τέτοιο προπολογισμό μακροπρόθεσμα κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο και γι' αυτό καλό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να μελετά την υπόθεση προς την κατεύθυνση αυτή. Ιδάλω την προσεχή φορά εγώ καταψηφίζω τέτοια μέσα προσωπικώς και παρεμποδίζω οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη. Τέτοιου είδους outsourcing, δηλαδή έξωθεν έλεγχος των ε, αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου δεν επιτρέπεται. γιατί είμαστε πλέον στο κιλό του κρεμου Και δεύτερον, μπορεί να υπάρχει μια πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των μέσων, όχι μόνο με την πρόσκληση κονδυλίων και από τα κράτη-μέλη και άλλους χορηγούς, αλλά και με την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των εφισταμένων μέσων του του προπολογισμού. Ναι, έστω, έτσι μας είπατε. Για να δούμε όμως τι, γίνεται, τι, θεωρείτε ότι γίνεται λάθος ε, ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τι λάθος κάνουμε ως προς την τήρηση των κανόνων του προϋπολογισμού ώστε τελικά να μην λειτουργεί το σύστημα όπως θα όφιλε να λειτουργεί. Δεν θα έπρεπε ο πρώτος κανόνας να είναι να ρυθμίσουμε ε, την τήρηση των κανόνων. Δεν θα πρέπει αυτό να συστήσουμε πρώτα απ' όλα. Η Επιτροπή λοιπόν και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού ασφαλώς θα πρέπει να ασχοληθούν εντατικά με την υπόθεση αυτή, ώστε να μην βρισκόμαστε διαρκώς σε μια τέτοια κατάσταση. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να διατυπώσουμε τροπολογίες ξεκάθαρες για να απευθυνθεί ένα σαφέστατο μήνυμα και προς την Επιτροπή και προς τα κράτη-μέλη. Αυτό και για το έκτακτο πακέτο για τα 9,2 δις και για όλα τα άλλα που ήμασταν διατεθειμένοι να βοηθήσουμε και να ε, σηκώσουμε μερίδιο του βάρους, αλλά δεν γίνεται ταυτόχρονα να ζούμε μία περίοδο κατά την οποία η καλή προαίρεση του Κοινοβουλίου ε, πέφτει θύμα καταχρήσεων και ε, παραγωνίστε το Κοινοβούλιο και οι αρμοδιότητες του δημοσιονομικές. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω την Αντιπρόεδρο κυρία Τζόρτζεβα. Την ευχαριστώ που ήρθε σήμερα εδώ. Φτάνετε και σε μια απόλυτος κατάλληλη στιγμή γιατί μιλούμε για ένα καταπίστευμα που ο κύριος Μπέγκε μας λέει ότι είναι ένα άθλιο εργαλείο το οποίο καταστρατηγεί τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το παραγωνίζει. Και απαιτείται η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου και προς την κατεύθυνση αυτή. Ο κύριος Δεπρέ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την ε, συνάδελφο Διαζαβάλ και τους ε, προευλαλήσαντες. Χρειάστηκε να δημιουργήσουμε με πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διαθέσή μας νέα έκτακτα χρηματοδοτικά μέσα. Υπάρχει το Μαντάτ, υπάρχει το ε, μέσο για το οποίο συζητάμε, υπάρχει το μέσο για την Τουρκία και φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και άλλα. Αυτό δείχνει τρία πράγματα κατά την άποψή μου. Το πρώτον, ότι τα όρια που είχε ορίσει το δημοσιονομικό, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο προφανώς δεν λειτουργούν, προφανώς δεν μας καλύπτουν γιατί καταλήγουμε να είμαστε υποχρεωμένοι να βρίσκουμε επιπλέον πόρους. Επομένω, έχουμε ένα μέρος του προπολογισμού να καλύπτεται από εθνικού πόρους. Δεύτερον, ότι οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του δημοσιονομικού πλαισίου είναι υπερβολικά αυστηροί και δεν μα δίνουν τη δυνατότητα να μετακινούμε κονδύλια για να αντιποκρινόμαστε σε έκτακτες ανάγκες. Και τρίτον, είναι ότι οι διαδικασίες που έχουμε για την χρήση των ε, κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι και αυτές υπερβολικά ε, γραφειοκρατικές και υπερβολικά αργές. Αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας στις ε, διαπραγματεύσεις για το μέλλον του δημοσιονομικού ε, πλαισίου. Πρώτον, τα ποσά, τα όρια και οι διαδικασίες για τη διάθεση των κονδύλιων. Γιατί αυτό που διαπιστώνουμε ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτό που λείπει από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό συμπληρώνεται από εθνικές πηγές, από τα κράτη-μέλη. Επίσης, δεν πιστεύω ότι στην ουσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χάνει τις εξουσίες της, τις αρμοδιότητές της, γιατί πάντοτε είναι επικεφαλής των ε, ε, διαφόρων επιτροπών που ε, διαχειρίζονται αυτά τα κονδύλια. Αλλά αυτό που στην πραγματικότητα γίνεται είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χάνει το ρόλο του, γιατί δεν, εξαιτίας αυτών των εκτάκτων διαδικασιών δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τη διάθεση του κονδύλιου. Είναι θέματα στα οποία θα επανέλθουμε όταν συζητηθεί το θέμα της αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου. Επίσης θέτει το θέμα της συνόδου της Βαλέτας. Είχε ε, λεχθεί ότι πρόκειται να χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένα έργα Συγκεκριμένε δράσει, λέει τον Εκκινοθέν, οι οποίες θα υποστηρίξουν την σταθερότητα στην περιοχή. Θα ήθελα να γνωρίσω ποιες είναι αυτές, τι έχει γίνει. Ο πρόεδρο θα κλείσουμε ε, και ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Μαλαγκάλ την συζήτηση εδώ, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Συμπερασματικά. Ακούσαμε την παρουσίαση της γνωμοδότησης. Είναι μια απειλή η οποία επικρέμεται, κυρία Αντιπρόεδρε, κάποια στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην ανέχεται πια αυτή την κατάσταση και να πει όχι και να αρνηθεί έναν προπολογισμό. Χρειάζεται λοιπόν να βρούμε έναν άλλον τρόπο στον οποίο τα κράτη-μέλη να δέχονται να συνεισφέρουν περισσότερα χρήματα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό με τι συνήθειε διαδικασίε, έτσι ώστε να μην παρακάμπτουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ανακοινώνω ότι οι τροπολογίες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι τις 5 Απριλίου 12 η ώρα. 26 Απριλίου θα συζητηθεί στην Επιτροπή και τις 4 Ιουλίου στην Ολομέλεια. Βλέπετε πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να υιοθετηθεί ένα μέσο το οποίο κατά τα άλλα το ονομάζουμε επίγον. Κύριε Κέιερ, μάλλον θα μπορούσατε να κάνετε μια σύντομη παρουσίαση για τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου. Ναι, πολύ σύντομα. Έχουμε ορίσει τη θέση μας το Συμβούλιο έχει ορίσει τη θέση του. Η Επιτροπή είπε ότι θα κοιτάξει να μας προσεγγίσει όσο περισσότερο γίνεται. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων έτσι, για εκείνο το απογευματάκι. Αυτά. Ε, donc, ε, Μάλιστα. Τριμερής διάλογος λοιπόν. Έγινε, έληξε. Θα ήταν ενδιαφέρον φαντάζομαι. Το ενδιαφέρον ήταν πάντως ότι το Συμβούλιο το εκπρούσε ο υπουργό των Οικονομικών των Κάτω Χωρών και σε αυτό είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Και τώρα ακούμε την κυρία Γεώργεβα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Χαίρομαι που μπόρεσα να παρακολουθήσω το τελευταίο κομμάτι της συζήτησης για το μέσον, για το καταπίστευμα για την ε, Τουρκία και θα ήθελα αν μου επιτρέπετε να κάνω κάποια σχόλια αμέσως πριν, πριν περάσουμε στην υπόλοιπη συζήτηση. Πρώτο σχόλιο. Είναι ευτύχημα για όλους μας, για την Ευρώπη, το Κοινοβούλιο επέμεινε στις διαπραγματεύσεις για το πολιετές νοσονομικό πλαίσιο ώστε να ανοίξει περισσότερο το περιθώριο της ευελιξίας, διότι αν δεν είχαμε την ευελιξία αυτή για την οποία επέμεινε το Κοινοβούλιο, θα βρισκόμασταν σε μια άκρος δύσκολη κατάσταση σήμερα. Το αναγνωρίζω αυτό και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο. Και βεβαίως θα πρέπει να αξιολογήσουμε, όπως είπε και ο κύριος Ντεπρέ, τον βαθμό επάρκειας αυτής της ευελιξίας και τι άλλο θα πρέπει ή θα μπορούσαμε να κάνουμε. Γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οι κλειδονισμοί είναι αλλεπάλληλοι, μερικές φορές και ταυτόχρονοι και χρειαζόμαστε μια ευελιξία την οποία ο παραδοσιακός ε, ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν διαθέτει. Δεύτερον, προσωπική μου δέσμευση είναι να εξασφαλίζεται η δημοκρατική ε, παλήθευση, εποπτεία και από τις δύο πλευρές της δημοσιονομικής ε, πτυχής. Ξέρω ότι υπήρχαν δυσφορίες σε σχέση με το καταπιστεύμα για την Τουρκία. Είχα την ευκαιρία εχθές να εξηγήσω την ε, διαδοχή γεγονότων που κατέστησαν το πρόβλημα κινητό στόχο και για την Επιτροπή που προσπαθούσε το δυνατό να κρατήσει ανοιχτό το θέμα, να ενημερώνει το κοινοβούλιο, αλλά με στόχο κινούμενο. Εν ώψη των πολλαπλών γύρων των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος Σούλτς, ήταν και στην Σύνοδο της Βαλέτα και σε κάθε Σύνοδο του Συμβουλίου. Βεβαίως, αναγνωρίζω ότι αυτό δεν υποκαθιστά δέσμευση διαρθρωμένη με το Κοινοβούλιο. Θα το πράξουμε. Θα το πράξουμε γιατί πια ο κόσμος είναι διαφορετικός και χρειάζονται μέσα διαφορετικά. Με τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση λοιπόν θα κοιτάξουμε να εξασφαλίσουμε συμμετοχή του Κοινοβουλίου, εμπλοκή του Κοινοβουλίου και για τέτοια μέσα, ώστε να λειτουργεί το σύστημα κατά τρόπο πλήρη και αποτελεσματικό. Φυσικά αυτό θα πρέπει και ταχύτητα να εξασφαλίσει και δυνατότητα αντιμετώπισης κινούμενων στόχων που προκύπτουν λόγω και της περιπλοκότητας των διαπραγματεύσεων, αλλά μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Και καθώς οι δικές μου προβλέψεις λένε ότι θα χρειαστεί να αναζητήσουμε τρόπους άντλησης σπόρων πολύ πιο βράχη πρόθεσμα για ε, απρόβλεπτες προτεραιότητες και αυτό σημαίνει και κονδύλια από τα κράτη-μέλη και μία δυνατότητα να δίνουμε απαντήσεις στα προβλήματα που αναδύονται. Η Γενική μας Διευθύντρια γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Και τώρα, επιτρέψτε μου να περάσω στο νέο μέσον κατεπίγουσας ενίσχυσης, ε, ε, βοήθειας. Πρόκειται για έναν τρόπο να ανταποκριθούμε σε ε, διαφορετικές και διαρκώς τροποποιούμενες ανάγκες και απαιτήσεις. Όπως ξέρετε παραδοσιακά, η ανθρωπιστική βοήθεια βλέπετε μόνο για τρίτες χώρες. Με εξαίρεση μία την Ιαπωνία μετά, τον, ε, μετά την καταστροφή της Φουκοσίμα το 2011. Κατά τα άλλα πρόκειται για χώρες φτωχές και αναπτυσσόμενες. Η μόνη πλούσια χώρα στην οποία προσφέραμε ανθρωπιστική βοήθεια ήταν η Ιαπωνία. Αλλά συζητούσαμε και είχαμε ήδη τη συζήτηση με μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοηθείας. Αυτό αποτελούσε ήδη ένα μήνυμα, το είχαμε δει δηλαδή ότι αποτελεί ένα μήνυμα πως ο κόσμος αλλάζει, αλλάζει ταχύτατα και βία και είναι πιθανόν μία πλούσια χώρα να βρεθεί ενώπιον τόσο μαζικών προβλημάτων που θα χρειαστεί ενίσχυση βοήθεια από αυτήν που παραδοσιακά προσφέρουμε σε αναπτυσσόμενες χώρες. Το να πράττουμε λοιπόν κάτι στο πλαίσιο της ε, προσφυγικής κρίσης σημαίνει ταυτόχρονα και είναι δική μου υπεποίθηση ότι χρειάζεται το μέσον διότι έχει αλλάξει ο κόσμος, διότι οι φυσικές καταστροφές, οι πλημμύρες, οι σεισμοί και το, είδαμε και στην ε, Ευρώπη αυτό αρκετέ φορέ, μπορούν να γονατίσουν ακόμη και την πιο πλούσια και οργανωμένη ε, εύρωστη οικονομικά χώρα και χώρα μέλος. Και γι' αυτό και τα νέα και το νέο αυτό μέσον κατεπίγουσας βοήθειας, παρότι συνιστά μια ε, άμεση αντίδραση σε αυτό που καθημερινά διαπιστώνουμε και αποτελεί επώδυνη υπενθύμηση αυτού νέου κόσμου στην Ελλάδα, αυτό που βλέπουμε η Ελλάδα έχει γονατίσει από το προσφυγικό. Ανταποκρινόμαστε λοιπόν στο συγκεκριμένο αυτό φαινόμενο, δημιουργώντας όμως ένα μέσον το οποίο θα μπορεί αντίστοιχα να αξιοποιηθεί για να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν αντίστοιχα απρόβλεπτες και σοβαρές συνέπειες και μέσα σε κράτος μέλος. Και με πολύ μεγάλη προσοχή μελετήσαμε τη νομική βάση του μέσου αυτού. Ε, εξετάσαμε διάφορα μέσα ε, άρθρα της συνθήκης το 214 συγκεκριμένα που είναι το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά το 214 ρητά αναφέρεται σε τρίτες χώρες. Άρα τρίτη χώρα μπορώ να πω ότι είναι η Ιαπωνία αλλά δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το 214 για την Ελλάδα για να σας το πω πολύ απλά. Κοιτάξαμε το μέσο για την πολιτική προστασία, το οποίο εγώ ιδιαίτερος υποστηρίζω και ξέρετε ότι ήμουν η Επίτροπος που το διαπραγματεύτηκε. Όμως η δυσκολία είναι προκειμένο, μάλιστα αυτό προβλέπει, η δυσκολία προκειμένου ότι προβλέπει μόνο ε, βοήθεια σε είδος. Είπαμε να αλλάξουμε το μέσον πολιτικής προστασίας ώστε να προσφέρει και οικονομική βοήθεια μέσω των οργανώσεων εταίρων μας. Καταλήξαμε όμως ότι δεν γίνεται αυτό. Λόγω της ανάγκης για ταχεία δράση. Είναι αποκεντρωμένη πολλές φορές η πολιτική προστασία σε πολλά κράτη-μέλη. Η αδίποτε λοιπόν αλλαγή θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να μπουν και τα, και τα γερμανικά λέντερ και οι, αντίστοιχα τα ομοσπονδιακά κρατήδια της Αυστρίας, ε, οι αποκεντρωμένες περιφέρειες της ε, Ισπανίας. Όλα αυτά λοιπόν δεν μας επέτρεπαν να αντιδράσουμε γρήγορα για να αντιμετωπίσουμε κατεπίψεις ανάγκες. Δηλαδή θα χρειαζόταν έως και χρόνια διαπραγματεύσεων. Με τη βάση αυτή λοιπόν, με δεδομένο αυτό, καταλήξαμε ότι το άρθρο που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση ήταν το 122 παράγραφος 1 που επιτρέπει να ληφθούν ταχαίως αποφάσεις όπως χρειάζεται και όπως χρειάζεται να οργανώσουμε τη δράση μας. Ωστόσο αυτό το άρθρο προβλέπει μόνο απόφαση από το Συμβούλιο και ξέρω ότι έχει γεννήσει πολλές ανησυχίες και αντιδράσεις σε επίπεδο κοινοβουλίου. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί. Ναι, το δημιουργούμε έτσι, αλλά ταυτόχρονα απευθύνουμε ένα σαφές μήνυμα στο κοινοβούλιο ότι ως δημοσιονομική αρχή θα επικυρώσει τις δημοσιονομικές συνέπειες αυτού του μέσου και οπωσδήποτε εμείς θα ενημερώνουμε και θα επιτρέπουμε την εμπλοκή σε όλη αυτή τη διαδικασία του Κοινοβουλίου εγκαίρως. Τι προτείνουμε σήμερα λοιπόν. και η απόφαση της Επιτροπής πέρασε χθε από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που την έκανε δεκτή. Προτείνουμε την ίδρυση αυτού του μέσου, τη σύσταση αυτού του μέσου για την αντίδραση σε κατεπίγουσες ε, συνθήκες ε, όπου χρειάζεται κατεπίγουσα δράση σε ενα ή περισσότερα κράτη-μέλη για λόγους ανθρωπιστικής υποστήριξης και όταν δεν προβλέπει κανένα άλλο μέσον τη δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες. 300 εκατομμύρια για το 2016. 200 για το 2017 και το 2018. Ο κύριος Φεράντες πολύ σωστά είπε μετά, μετά το 2018. Ελπίζουμε ότι θα εξαλειφθεί ο λόγος ύπαρξής του. Αν και η πρόβλεψή μου είναι προς το αντίθετο. Εν πάση περιπτώσει τώρα πρόκειται για αντίδραση στην προσφυγική κρίση. Ελπίζουμε σε τρία χρόνια να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και έτσι το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα να μην είναι τόσο οξύ. Και έτσι μέχρι τότε θα έχουμε μπορέσει να οργανώσουμε πιο σωστά μια φόρμουλα για το μέλλον, χωρίς να θέλω σήμερα να προδικάσω το τι θα προκύψει από την ε, συλλογική μελέτη και φρόνιμη απόφαση που θα προκύψει στη συνέχεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να θεσπιστεί μια ε, γραμμή προϋπολογισμού για τα πρώτα 100 που θα είναι ε, η προκαταβολή από το ΆΜΙΦ 100 εκατομμύρια θα πάρουμε όπου ξέρουμε ότι υπάρχουν 400 εκατομμύρια για την επανεγκατάσταση. Ξέρουμε ότι το, έργο, το σχέδιο αυτό επανεγκατάστασης δεν θα μπορέσει να απορροφήσει τους προσεχείς 6 μήνες, 7-8 μήνες το ποσό αυτό που έχει προβλεφθεί και άρα μπορούμε να αντλήσουμε από εκεί ποσά. Ο κύριος Γκάιερ ρωτούσε τι έγινε, αλλά τελικά ρωτάει κιόλας εάν αρκούν τα ποσά. Η δική μας πρώτη εκτίμηση είναι ότι πρέπει να το κοιτάξουμε, να δούμε στο τρίτο ή και στο τέταρτο κεφάλαιο, εφόσον από εκεί έχουν εξαντληθεί τα ποσά και δεν υπάρχουν περιθώρια, γιατί θα φτάσουμε στο σημείο αυτό, αλλά δεν θέλουμε να προδικάσουμε την κατάσταση πριν φτάσει η ώρα να το δούμε έτσι. Επίσης, προτείνουμε να δοθούν στη Europol οι απαραίτητοι πόροι για ένα κέντρο, υποδοχή, ένα κέντρο ελέγχου. Ξέρω ότι αυτό το υποστηρίζει το, το Κοινοβούλιο. Και αυτό έχω έρθει να σας προτείνω. Σύντομα, η λογική, η, ο συλλογισμός πίσω από τη δημιουργία αυτού του μέσου κατεπίγουσας βοήθεια και ο συλλογισμός πίσω από την επιλογή της νομικής βάσης, πρώτον. Δεύτερον, διευθέτηση και συμφωνίες περί χρηματοδότησης και τρίτον, δεδομένου ότι είμαι και εδώ αναφέρω και το θέμα της Europol και τις ανάγκες της Europol απολύτως αιτιολογημένες και στις οποίες μπορούμε να ανταποκριθούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Αντιπρόεδρε για αυτή την αναλυτική παρουσίαση. Είναι σίγουρο ότι δεν έχετε εύκολο έργο. δεδομένων των συνθήκων που είναι τραγικές. Χρειάζεται λοιπόν να σκεφτούμε όλοι μαζί και η αναθεώρηση του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Μήπως αντί να δημιουργούμε αυτά τα κατεπιστευματικά ταμεία και αυτά τα ε, επιπλέον ταμεία, να δημιουργήσουμε ένα ε, ταμείο το οποίο θα μπορούσε να ε, χρηματοδοτεί κρατημέλη που χρειάζονται να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις, παραμένοντας όμως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Κύριε Φερνάντες. Σας ευχαριστώ. Καλώς ορίζω την Επίτροπο. Συμφωνώ μαζί σας κύριε Πρόεδρε ότι δεν έχει εύκολο έργο μπροστά της κυρία Γεωργίεδα. Εκείνη θα πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις ικανότητες και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας για να λύσουμε την ανθρωπιστική κρίση που υπάρχει πλέον εντός των σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε εδώ μια περίπτωση όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δράσει γρήγορα. Δύο ημέρες πριν, μόλις, συζητούσαμε την μεταφορά ε, κονδυλίων 5 εκατομμυρίων ευρώ στο ε, του Ταμείου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και να από δύο μέρες μετά το θέμα θα τεθεί ξανασυζητάτε. Δεν ξέρω πώς τελικά θα την ονομάσουμε αυτή τη μεταφορά κονδυλίων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δείχνει ότι όταν χρειάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιποκριθεί γρήγορα, το κάνει. Τώρα όσον αφορά αυτό το νέο χρηματοδοτικό μέσο, νομίζω είναι προφανές ότι θα το εγκρίνουμε, γιατί υπάρχει μια επίγουσα ανάγκη. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι αυτή την ανάγκη την επίγουσα θα μπορούσαμε να την είχαμε προβλέψει. Και οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μας ρωτήσουν κάποια στιγμή. Πώς γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκρίνεται τόσο γρήγορα όταν έχουμε προβλήματα εκτός των συνόρων της και να καθυστερεί τόσο χαρακτηριστικά όταν τα προβλήματα βρίσκονται εντός των συνόρων της. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που θα μας ρωτήσουν. Ένα άλλο ερώτημα που εμένα με ε, προβληματίζει είναι ότι αυτό το χρηματοδοτικό μέσο δεν προβλέπεται για τους πρόσφυγες και ε, μόνο, αλλά για οποιονδήποτε άλλον εντό των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να βρεθεί και βρίσκεται σε μια έκτακτη ανάγκη αντίστοιχη με αυτήν των προσφύγων σήμερα. Επομένως, κατά την άποψή μου δεν έχει νόημα να θεωρούμε ότι το μέσο αυτό μπορεί να μην ε, είναι μόνιμο, να μην το εντάξουμε στο πλαίσιο του γενικού προπολογισμού, σαν να μην ήταν, ε, σαν να μην ήταν ε, η, η ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια εντός των συνόρων κάτι που θα συνεχίσει να υπάρχει στα επόμενα χρόνια. Είναι μια έκτακτη ανάγκη που είναι εξαιρετικά οξία η κατάσταση σήμερα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα εξαλειφθεί το 2018 ή 2019. επομένω. αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο δεν θα μπλοκάρει αυτή την πρωτοβουλία, αλλά ε, θα απευθύνει μια έκκληση προς την Επιτροπή ε, να ε, φροντίσει έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μην περιθωριοποιηθεί. Το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί την ε, εκτέλεση του προπολογισμού, τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Δεν πρόκειται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πεμπολίσει των αρμοδιοτήτων του με τόση ευκολία και με τόση καλή θέληση. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μια έκτακτη κατάσταση, την οποία όμως θα μπορούσαμε να είχαμε προβλέψει. Αναγνωρίζω όμως ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και ότι έχει επιδεινωθεί από το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, δεν έχουν υλοποιήσει τις υποσχέσεις που είχαν δώσει. Το οποίο μας καταδεικνύει ότι θα είχαμε μια επιπλέον εξασφάλιση, μια επιπλέον εγγύηση αν γνωρίζαμε ότι χρησιμοποιείται η διαδικασία του ευρωπαϊκού προπολογισμού για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνουμε. Θα εγκρίνουμε λοιπόν τη δημιουργία αυτού του μέσου τροποποιώντας τον, το δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά βέβαια υπάρχουν οι διαδικασίες. Το οποίο σημαίνει ότι αυτή η, τροποποίηση του προπολογισμού θα πρέπει να γίνει ένα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Δεν μπορεί να γίνει κάτι πιο νωρίς. Και αυτό τι μας δείχνει, ότι αν είχαμε ένα ειδικό μέσο το οποίο θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε οποτεδήποτε προκύπτει μια επίγουσα ανθρωπιστική ανάγκη, που να προβλέπεται το δημοσιονομικό πολιτεύθυνο το δημοσιονομικό πλαίσιο, που να υπάρχουν σχετικέ διαδικασίε, που να επιτρέπουν οι σχετικέ διαδικασίε να χρησιμοποιείται γρήγορα, δεν θα χρειαζόταν να περιμένουμε την ολομέλεια του Απριλίου. Γιατί εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Απ' τη μία λέμε ότι αντιποκρινόμαστε σε μια εκτακτή ανάγκη, απ' την άλλη λέμε ναι, αλλά πρέπει να περιμένουμε την, ολομέλεια του, τη μικρή ολομέλεια του Απριλίου πόσο πιστικοί μπορούμε να είμαστε ενώπιον των πολιτών όταν τα λέμε αυτά τα δύο ταυτόχρονα. Χρειάζεται να έχουμε γρήγορες ε, απαντήσεις σε επίγοντα προβλήματα. Ευχαριστώ πρόεδρε να είμαι σύντομη μια που ο κύριος ε, Φερνάντες με όσα είπε κάλυψε βεβαίω κυρία Επίτροπε πρόκειται να βοηθήσουμε και να υπάρξει μια τέτοια ανθρωπιστική βοήθεια και εδώ στην Ένωση είναι κατεπήγον το θέμα όπως έλεγε ο κύριος Φερνάνδε για τα πράγματα φαινόντουσαν προς τα που πάνε δυστυχώς χρειάζεται ένα τέτοιο μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα στα σύνορα της Ένωσης και κατεπηγόντως θα πρέπει να το θεσπίσουμε αυτό το μέσο, να μαζέψουμε αυτά τα πρώτα εκατομμύρια ε, από το ΑΜΙΦ έχουμε κάποια κονδύλια, αλλά βέβαια ε, δεν μας αρέσουν τέτοιες διαπραγματεύσεις γιατί όταν έχουμε νέα ταμεία να έχουμε και καινούργια κονδύλια αλλά γνωρίζουμε ότι όταν κάτι επήγει θα πρέπει να επιστρατευτούν τα υπάρχοντα χρήματα. Βεβαίως και είναι πάρα πολύ στενάχωρο το ότι έχουμε αυτά τα χρήματα στο ΑΜΕΦ και τώρα θα πρέπει να τα εκταμιεύσουμε ε, για αυτή την ε, πολιτική για το προσφυγικό. Δεν φταίει ούτε η Κομισιόν ούτε βέβαια το Κοινοβούλιο. Ε, φταίει αυτή η θλιβερή στάση των κρατών μελών που για το προσφυγικό αναζητούμε τώρα ε, χρηματοδότηση. Οπότε και εγώ από πλευράς των Σοσιαδημοκρατών συμφωνώ με αυτό το καινούριο χρηματοδοτικό μέσο να προσέξουμε όμως να υπάρξει πρικοδότηση και να χρησιμοποιηθούν ιδέουσες διαδικασίες. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Τόμα. έχετε το λόγο. Με ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Σίγουρα. Και έχουμε επίγνωση του κατεπήγοντος. Δεν έχω καμία διάθεση αμφισβήτησης. του αντίθετο θα υποστηρίξουμε. Όλα αυτά διαπιστώνεται όπως και εμείς ότι έχουμε ξεκινήσει μια πορεία για την άξιση του προϋπολογισμού που είναι όλο ένα και πιο δύσκολη. Ε, δεν λέω ότι άνθουν τα δημοσιονομικά τον αντίθετο εδώ και κάποια χρόνια. Πάντως ε, το, τα κατεπήγοντα απαιτούν και κατεπήγουσες λύσεις. Οπότε ε, το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας. Ούτε έχει την ουδέουσα ευελιξία. Ούτε καν έχει τις απαραίτητες οροφές που απαιτούν οι κατεπίγουσες περιστάσεις. Ακούσατε, από τον κυρία Καρδιά Θάμπαλ, από τον κύριο Μπέγκε, από τον κύριο Ντεπρέ, ότι όσον αφορά το μέσο χρηματοδοτιστής της Τουρκίας, εμείς θεωρούμε ότι εδώ υπάρχει κάτι σαν κορεσμός ε, πέραν του κατεπίγοντος, γιατί κάθε φορά αυτά τα οποία θεσπίζουμε αφορούν το εξωτερικό της Ένωσης. Χρειάζεται περισσότερο περιθώριο λιγμών. Κανείς δεν το λέει. Αλλά είπαμε ότι είναι κατάσταση κατεπίγουσα και εγώ καταλήγω στο ότι ήρθε η ώρα αυτά τα στοιχεία να τα λάβουμε υπόψη για μια αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Και όπως είπε και ο πρόεδρός μας, και εγώ είμαι υπέρ, να έχουμε κάποιο είδους αποθεματικό για τα κατεπήγοντα, το οποίο να διακρίνεται από ευελιξία και ακριβώς σε περίπτωση κατεπήγοντος να έχει αυτή την δέουσα ε, ευελιξία, αλλά να είναι στα πλαίσια του κοινοτικού προϋπολογισμού, να επιδέχεται ε, τον εκ των έλεγχο, με τους πιο ευέλικτους δικούς μας ε, κανονισμούς και διαδικασίες. Και εδώ μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό στην Επιτροπή μας. Για αυτή την αναθεώρηση να μας πείτε πώς το βλέπετε. Τι χρονοδιάγραμμα βλέπετε εσείς για την αναθεώρηση του μεσονομικό πλαίσιο. Ο πρόεδρος δίνει το λόγο στον κύριο Ντεπρέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και πολύ σύντομα. Εγώ και η ομάδα μου συμφωνούμε πολύ με την πρωτοβουλία αυτή. Νομίζω ότι αισθανόμαστε όλοι ντροπή που αφήσαμε την Ελλάδα ε, να αντιμετωπίζει μια μαζική ροή ε, προσφύγων για τόσο καιρό δεδομένων των οικονομικών δυσχεριών στις οποίες βρίσκεται. Για τα πρόστα κονδύλια για το Europol δεν συζητήσαμε ούτε για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Όντας Βέλγος, οφείλω να πω, πρέπει να κοιτάμε και αυτά που γίνονται σήμερα στις Βρυξέλλες. Οι κίνδυνοι δεν είναι στο παρελθόν, δεν ανήκουν στο παρελθόν. Ενδέχεται να υπάρχουν ακόμα σοβαροί κίνδυνοι μπροστά μας. Για την πρότασή σας, συμφωνώ απόλυτος με την πρόταση και σημειώνω με ενδιαφέρον πως προτείνετε τη δημιουργία ενός νέου κεφαλαίου στο κεφάλαιο 3. Χαίρομαι που μπορεί να υπάρξει ένα νέο κεφάλαιο, γιατί έτσι μπορούμε και όταν έρθει η ώρα για την αναθεώρηση του του οικονομικού πλαισίου να υποστηρίξουμε την πρόταση μιας διαρθρωμένης ανατροφοδότησης. Ξέρω ότι αρκετοί το έθιξαν ήδη, θα είναι ενδιαφέρον όμως και χρήσιμο αυτό για την διαπραγμάτευση. Η σύντομη φράση που περιλαμβάνεται στο κείμενο που αναφέρεται ότι θεωρείται πρόωρο, υπογραμμίζω, πρόωρο προς το παρόν, την την αξιοποίηση του contingency margin, του ε, περιθωρίου έκτακτη ανάγκης. Το λέτε πρόωρο, άρα δεν αποκλείεται στο μέλλον να αξιοποιηθεί. Επίση, επιτρέψτε μου για την διαχείριση αυτή τη πρωτοβουλία ε, να σα πω ότι έχουμε κάποιε επιφυλάξει σχέση με τι θέσει εργασία που θα χρειαστούν και που θα αναδιπλωθούν σε σχέση με δράσει τη αστυνομία που έχουν να κάνουν κατά τα άλλα με την ασφάλεια. Με ξαφνιάζει αυτό ή μη τι άλλο πρέπει να το πω. Έχουμε θέματα προτεραιότητα της ασφάλειας, για την ε, χρηματοδότηση του προσωπικού αυτής της νέας πρωτοβουλίας. Παίρνουμε λεφτά από το Ταμείο Ενίσχυσης των Μέσων για την ε, ασφάλεια. Δεν καταλαβαίνω. Παράδοξο μου φαίνεται. Ή μη τι άλλο. Τελευταίο σημείο. Όπως και ο κύριος Φερνάντες. Για τα κατεπήγοντα. Νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσουν θέματα και προτιμήσεων στα κράτη που μπορούν να οδηγήσουν σε πιο σύντομες διαδικασίες. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να δεχθούμε μονίμως να μας πιέζουν διορίες που δεν είχαν ε, θεσπιστεί για να, για να αντιμετωπιστούν τέτοια κατεπήγοντα ζητήματα. κύριος Μαραγάλ. Πρόεδρε, να μην επαναλάβω αυτά το οποίο ελέγχθησαν. Έτσι κι αλλιώς συμφωνώ και για το περιεχόμενο, όσον ακούσαμε και για το περιεχόμενο ε, αυτού του καινούργιου μέσου και συμφωνώ ότι είναι κάτι επίπεδο. Αλλά, για να δούμε ευρύτερα το θέμα. Το θέμα δεν είναι αν θα καινοτομήσουμε δημιουργικά, αλλά το τι πολιτική θα καλύψουμε με αυτή την καινοτομία. να δούμε τι θα κάνουμε σε σχέση με αυτό το χρηματοδοτικό μέσο προς την Τουρκία. Τι έχουμε, έχουμε τρία δις, συν άλλα τρία δις. Αυτό δεν λέμε. Και πριν λέγαμε για αυτό το ευρωπαϊκό κατάπίστευμα, το οποίο είπαμε ότι ο πλευρά χρηματοδοτικής διαχείρισης είναι μια καινοτομία και είπαμε ότι δεν δικαιολογείται 100% για μας γιατί μας βγάζει από το παιχνίδι κάπως. Δεν θα έχουμε τον έλεγχο. Αλλά την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε ε, κατά πόσον θα θυσιαστούμε για να βάλουν τα κράτη-μέλη αυτά τα χρήματα. Πάντως δεν είναι και τόσα πολλά τα λεφτά που θα βάλουν τα κράτη-μέλη τόσο ώστε να δικαιολογήσουν αυτή την εγκατάλειψη. Δεν είναι αρκετή αυτή η πρικοδότηση. Όπω ελέγχθη σωστά, πρόκειται για μια αναδιόρεση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό και γίνεται. Άρα, το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο το που πάμε. Όμως, έμεσα προκύπτει από μια ανησυχία. Άρα είπαμε ότι δίνουμε τα 3 δις για να μην έρθουν εδώ οι πρόσφυγες. Και είπαμε 700 εκατομμύρια για να μην βγουν οι πρόσφυγες από την Ελλάδα. Μα αν εκεί θέλουμε πάνε τα χρήματα τότε δεν συμφωνώ. Ή θα πρέπει να καλύψουμε όλη την Ευρώπη για την κατάσταση ανάγκες, για την μετεγκατάσταση κλπ. η κίνηση δεν έχει νόημα. Οπότε και εγώ διαφωνώ. Εάν πρόκειται να εξυπηρετήσει για μια πολιτική ε, περιορισμού, ε, από τη μια μεριά περιορισμού στην Τουρκία και περιορισμού των, του, του, ροών στην Ελλάδα, τότε. Γιατί αυτό δεν είναι θέμα κατεπίγοντος. Δεν μπορεί αυτό το, το καινούργιο μέσο χρηματοδότησης να έχει αυτό το σκοπό. Άσχολτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σύντομα θα πω ότι η ομάδα μου θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία αυτή. Έχουμε γνώση του γεγονότο ότι η Επιτροπή ανταποκρίνεται σε μια κρίση. Μια κρίση όπου οι τρέχουσε δομέ είναι ε, ακατάλληλε για να αντιμετωπίσουν. Πρώτον λοιπόν, θα συμφωνήσω με, την, ε, με τα σχόλια των συναδέλφων προς την ανάγκη για ταχύτατη δράση. Δεύτερον, για να ζητήσω να με διαβεβαιώσετε ότι υπάρχει όντως η δυνατότητα απορρόφησης των κονδυλίων αυτών. Υφίστανται οι απαραίτητες υποδομές σε παραδείγματι. Γιατί πολύ συχνά παρατηρούμε ότι μπορεί με τις καλύτερες προθέσεις να στέλνουμε χρήματα, αλλά να μην είναι το ίδιο πράγμα με χρήματα που αποτελεσματικά δαπανώνται. Ολβρίχτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συμφωνήσω με τα σχόλια της κυρίας Τωμά η ε, εισηγήτη της για την αναθεώρηση και να σημειώσω ότι αυτό που κάνουμε τώρα αναθεώρηση είναι. Και όχι σήμερα. Από την πρώτη στιγμή άρχισαμε να αλλάζουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Από την αρχή ακολουθούμε κανόνες άλλους από αυτούς του MFF. Λοιπόν, καλό θα ήταν πρώτα να κοιτάξουμε, να συνοψίσουμε ότι έχουμε ήδη αλλάξει σχέση με τον κανονισμό του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, γιατί είναι ξεκάθαρο στον κανονισμό ότι χρειάζεται να διαφυλαχθεί η ενότητα του προϋπολογισμού. Πρώτο ερώτημα λοιπόν, αυτό είναι ενότητα του προϋπολογισμού. Συνεργάζονται τα όργανα ή μήπω τελικά συζητούμε όχι μόνο τον προϋπολογισμό, όχι, όχι τον προϋπολογισμό μόνο, αλλά ολόκληρο το σύστημα, το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί περί αυτού πρόκειται. Έχουμε λοιπόν δύο προϋπολογισμούς, αυτών των οποίων ορίζουμε με σταθερά στοιχεία και των οποίων ε, συνδέουμε με προτεραιότητες και θα, έχει μια διάρκεια 5 ή 10 ετών και έναν άλλον προϋπολογισμό που θα ας το πούμε και αυτόν τον προπολογισμό, όπου τα κράτη-μέλη θα αποφασίζουν πως αν συμβεί κάτι θα ρίχνουν χρήμα και άρα θα ορίζουν νέες προτεραιότητες που όμω είναι προτεραιότητα όχι μόνο των κρατών μελών αλλά και ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου και ποια είναι η αναλογία μεταξύ του πρώτη κατηγορία προπολογισμού και του έτερου. 90% ο πρώτος, 10% άλλος και σταδιακά θα πάμε στο 40-40-50-50, 40-60-50-50. Η συζήτηση για την αναθεώρηση νομίζω ότι γίνεται όλο και πιο σοβαρή. Δεν υπάρχει εμβόλιο ότι χρειάζεται αυτό που συζητούμε σήμερα. Κανείς δεν θέλει να το παρεμποδίσει. Είναι απαραίτητο, αλλά η σημερινή απόφαση ταυτόχρονα επηρεάζει και τις αυριανές αποφάσεις. Ό,τι κάνουμε σήμερα που αποφασίζει και επηρεάζει τις επιλογές του αύριο, τι θα γίνει με τις δομές σε δύο χρόνια. Γιατί να μην υπάρξει αποθεματικό, γιατί να μην συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη και θα θυμάστε ασφαλώς τις δραστηριότητες του κυρίου Λεβαντόφσκι όταν τον είχαμε ρωτήσει πόσα χρειαζόμαστε για τις δομές 2020 για να διαπιστώσουμε, για τη στρατηγική 2020, για να διαπιστώσουμε ταχύτατα ότι δεν υπήρχαν χρήματα για τη στρατηγική 2020. Άρα να πούν τα κράτη-μέλη τι θέλουν, τι προτεραιότητες έχουν, πόσο θα κοστίσει αυτό και τι αποθεματικό προβλέπουν. Αποθεματικό για κατεπίγουσα ανάγκη, ειδικέ ανάγκες, ό,τι θέλετε. Ή αλλιώς ορίζουμε τις προτεραιότητες και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε αναλόγως. Πολιτική ερώτηση που θα κρίνεται πολιτικά και στις χώρες μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της ε, ειδική μου, τι θα κάνουμε τα χρήματα, προσδιορίζουμε ένα αποθεματικό ή ζητάμε κάθε δύο-τρεις μήνες από τα κράτη-μέλη περισσότερα χρήματα για συγκεκριμένους στόχους. Γιατί θα ρωτάει ο κόσμος πόσα ακόμα θα δώσουμε και θα ξαναδώσουμε και θα ξαναματαδώσουμε. Κατεπίγουσα ανάγκη, μα δεν πρόκειται για κατεπίγουσα ανάγκη πλέον, πρόκειται για αλλαγή συστήματος. Ενό συστήματος που στηρίζεται σε προσωρινές λύσεις και όπου η Επιτροπή δεν είναι πλέον φορέας δράσης, αλλά υπηρεσία διαχείρισης. Ο Πρόεδρος. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο, επομένως κυρία Αντιπρόεδρε. Συμφωνούμε όλοι ότι έχετε ένα δύσκολο έργο. Το αναγνωρίζουμε, σας εκτιμούμε και προσωπικά και για το έργο σας. Ωστόσο εδώ βρισκόμαστε στην Επιτροπή Προπολογισμού. Έχουμε κλειδιά από του Ευρωπαίους πολίτες. Προσπαθούμε το έργο μας να είναι ορθό και κατανοητό. Πρέπει να μπορούμε να εξηγούμε στους πολίτες τι κάνουμε και ποιος είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που γίνεται είναι πλήρως ακατανόητο. Α, σαν να βρισκόμασταν κάπου μακριά σε μια γυάλα και ο λαός να μην καταλάβει. Έχουμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα συνήθεια και κάθε φορά που υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη θα ψάχνουμε επιπλέον χρηματοδότηση, επιπλέον κονδύλια. Μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Το ερώτημα είναι αν η αρχή των ε, κρατών μελών και οι υπουργοί οικονομικών τους έχουν ε, θέσει αυτό το θέμα, έχουν συζητήσει αυτό το θέμα. Προβλέπεται η αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και γνωρίζουμε ότι αυτό θα δημιουργήσει σύγκρουση. Αλλά τι μπορούμε εμείς να ζητήσουμε και να τους πούμε από την πλευρά μας έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ενότητα του προπολογισμού. Βεβαίως, ο κ. Γιούνκερ μίλησε για έκτακτες καταστάσεις, επομένως χρειάζονται και έκτακτοι πόροι. Δεν θα είναι απλό. Αλλά χρειάζεται και ένα πλαίσιο. Γιατί διαφορετικά το σύστημα που δημιουργούμε γίνεται όλο και πιο παράλογο και κάποια στιγμή δεν θα λειτουργεί. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας και αν θέλετε έχετε το λόγο παρακαλώ. Thank you very much for the comments that have been made. I understand you have Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που μου απευθύνατε. Γνωρίζω ότι έχετε φορτωμένη η ημερησία διάταξη, επομένως θα προσπαθήσω σύντομα να απαντήσω. Λοιπόν, πρώτον, αν αλλάζει ο προπολογισμό, χρειάζεται. Αυτό είναι ε, μια πραγματικότητα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονό ότι στο παρελθόν είχαμε μια ισορροπία ανάμεσα σε εκείνους που ήθελαν τους αγροτικούς πόρους, τα ταμεία συνοχής και το rebate και είχαμε βρει μια ισορροπία. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η ισορροπία δεν λειτουργεί πλέον. Φαίνεται ότι αυτή η δημοσιονομική ειρήνευση που είχαμε επιτύχει δεν θα λειτουργεί πια. Και σιγά σιγά δημιουργεί ένα κόστος που δεν θέλουμε να αναλάβουμε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά που απασχολούν και ενησυχούν τους πολίτες μας. Και είμαι περήφανη για αυτό που καταφέραμε, γιατί καταφέραμε να διαθέσουμε 6 δισεκατομμύρια ευρώ ε, πολύ γρήγορα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την εκτακτή κατάσταση. Δεν ήμουν παρούσα στην προηγούμενη συζήτηση, αλλά ε, ρωτάει ο κόσμος τι κάνετε. Να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Ε, στην Τουρκία υπάρχουν ήδη δύο έργα. Πρώτον, 140.000 παιδιά από τη Συρία πηγαίνουν στο σχολείο το οποίο γνωρίζουμε ότι επίσης ότι από τη στιγμή που τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο η πιθανότητα η οικογένειά τους να προσπαθήσει να πάει αλλού μειώνεται και επίσης έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα με κουπόνια, με μια κάρτα μάλλον, ηλεκτρονική, για να μπορούν να αγοράζουν οι πρόσφυγες ε, τα τρόφιμα τους και τα είδη πρώτης ανάγκης. περίπου 40.000 ε, πρόσφυγες καλύπτουμε με αυτόν τον τρόπο και πάλι μειώνεται η πιθανότητα αυτοί οι πρόσφυγες να αποφασίσουν να μετακινηθούν. Επομένως, δεν ρίχνουμε χρήματα αλόγιστα, προσπαθούμε να βρούμε ε, λύσεις σε μία κατάσταση είναι ξεκάθαρο ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τις μαζικές αφήξεις προσφύγων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από καμία χώρα μόνη της. Πέντε εκατομμύρια πρόσφυγες φεύγουν από τη Συρία οπουδήποτε και να πάνε θα δημιουργηθεί ένα, ε, ένα σοκ. Αλλά θα πρέπει και εμείς να προετοιμαστούμε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του προπολογισμού να απαντήσουμε στις δύσκολες ερωτήσεις που μας θέτουν οι πολίτες μας. Το ζήτημα δεν είναι να δίνουμε μάχες άνευ αλλά να συνεργαστούμε για να απαντήσουμε στα πραγματικά προβλήματα μέσα στο πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Πρώτα απ' όλα ότι χρειάζεται να υπάρχει ομοφωνία, έτσι έχουν τα πράγματα, και επίσης στο γεγονό ότι έχουν υπάρξει κάποιε συμφωνίε στο παρελθόν που δεν υπάρχει περίπτωση τουλάχιστον δεν μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα υπάρξει ομοφωνία να αλλάξουν. Πρέπει να δούμε λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο τι μπορούμε να κάνουμε, να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που έχουμε για να καταλήξουμε σε καλύτερη διάθεση των ε, κοντιλίων του προπολογισμού. Γι' αυτό εμείς θα προσπαθήσουμε. Συμφωνώ με εκείνους που είπαν ότι την έκτακτη αυτή ανάγκη μπορούσαμε να την είχαμε προβλέψει. Δύο χρόνια πριν τα έλεγα αυτά και τώρα δεν ε, χαίρομαι που διαπιστώνω ότι είχα δίκιο. Δεν επιχαίρω, αλλά γνωρίζαμε ποια είναι η κατάσταση και επιλέξαμε να εθελετυφλούμε μέχρι που δεν μπορούσαμε πια να την αγνοήσουμε γιατί έφτασε στην πόρτα μας. Είναι όπως τον καπνιστή που αποφασίζει να κόψει το κάπνισμα όταν έχει πάθει πια καρκίνο του πνεύμονα και δεν έχει νόημα. Δεν το λέω αυτό για να μας δικαιολογήσω, αλλά όταν εξελισσόταν η κρίση με την οικονομία της Ελλάδας, Ήδη τότε συζητούσαμε στην Κομισιόν εάν χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ε, χρηματοδοτικό μέσο για την ανθρωπιστική βοήθεια εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιατί ήδη λέγαμε ότι μπορεί να χρειαστεί. Και οι αντιδράσει ήταν μα γιατί δεν υπάρχει περίπτωση η Ευρώπη είναι δυνατή, είναι ισχυρή, δεν θα το χρειαστούμε ποτέ αυτό το πράγμα. Και δέχομαι να μου ασκήσει κάποιο κριτική, θα έπρεπε να είχα επιμείνει περισσότερο τότε. Τώρα κάτι έχουμε παρόμοιο ε, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα ένα δίκτυο 200 οργανώσεων για την παροχή ανθρωπιστικής ε, βοήθειας εκτός ε, ένωσης. Ήδη μιλάμε με την Διεθνή Επιτροπή Αριθμού Σταυρού, με την Υπατερμοστία του για τους πρόσφυγες, με το Save the Children, με τη UNICEF, με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται επί τόπου, ελληνικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις όπως η Αλληλεγγύη, που έχουν γνώση της κατάστασης. Και παρεπιπτόντως πριν την Ολομέλεια του Απριλίου γνωρίζω επειδή αυτές οι οργανώσεις μας εμπιστεύονται θα, ξεκινήσουν να δαπανούν χρήματα προσβλέποντας ε, ε, στα χρήματα που θα τους έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη βοηθούν ελπίζοντας στους πόρους που θα έρθουν. Προσωπικά θα ε, προσπαθήσω να βρω ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο για να εμπλέκεται το Κοινοβούλιο στον έλεγχο της διάθεσης των κονδυλίων αυτών των χρηματοδοτικών μέσων. Γιατί η κρίση υπάρχει και πρέπει να βρούμε τρόπους για να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που δεν είχαμε προβλέψει με την εμπλοκή του Κοινοβουλίου. Όλοι γνωρίζουν ότι και στους εθνικούς προϋπολογισμούς υπάρχουν ειδικοί λογαριασμοί για έκτακτες καταστάσεις. Αλλά στα κράτη, το εθνικά κοινοβούλια πάντα ελέγχουν την εκτέλεση αυτών των προϋπολογισμών. Και τώρα που άλλαξε ο κόσμος θα πρέπει και εμείς να επινοήσουμε το πώς θα τις καλύψουμε και να υπάρχει το δικαίωμα του ελέγχου. Κάτσαμε και τα συζητήσαμε, βρήκαμε την απάντηση και αυτό και θα κάνουμε εμείς επίσης τέλος. Ε, θα πρέπει να είστε περήφανοι για το εξής. Λέτε ότι χρειάζεται περισσότερη ευελιξία. Ε, ναι. Εσείς το καταφέρατε. Το ότι κάνουμε κάτι εσείς το καταφέρατε κι άρα. Αυτό το μήνυμα θέλω να στείλω στο Κοινοβούλιο ότι εσείς καταφέρατε να γίνει αυτό με τον προϋπολογισμό και ελπίζω να αισθάνεστε περήφανοι γι' αυτό. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Γενική Συγητά, Θέλετε το λόγο. Φέροντες. Συντομότατα να σας πω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ενεργούμε ταχύες όταν πρόκειται περί επίγοντος, παίρνουμε τα χρήματα από την ανθρωπιστική βοήθεια και γίνεται αυτή η μεταφορά πόρων για τους πρόσφυγες. Μας το πριν από δύο μέρες και δεν το κάνουμε σήμερα. Και επίση όσον αφορά αυτόν τον αγώνα είμαστε στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί θυμάμαι επίση ότι σε κάποιες συναντήσεις μας δυσκολευτήκαμε πολύ για να βρούμε ευελιξία για τον προϋπολογισμό του 16. Χωρίς την ευελιξία αυτή η κατάσταση θα ήταν χαοτική αλλά όλες οι πολιτικές ομάδες, όλο το κοινοβούλιο ε, ποντάρουν πάνω σας. Ωραία. Επομένω, με αγωνία περιμένουμε ε, στις 4 Απριλίου την ε, γνωμοδότηση του κ. Φερναντές και αυτή η έκθεση θα ψηφιστεί στις 11 Τετάρτου και 13 ή 14 θα την κατεβάσουμε στην Ολομέλεια. Και πάλι ευχαριστούμε κυρία Αντιπρόεδρε τη Επιτροπής. είμαστε στο πλευρό σα, αλληλέγγυοι, με θαυμασμό κλπ. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζει ο Πρόεδρος. Το σημείο υπάρχουν 5, είπαμε ότι δεν θα ζητηθεί τώρα όσον αφορά αυτέ τι ε, προπαρασκευαστικές δράσεις κλπ. για τη χρήση 16-17. Οπότε τώρα, αυτά τα πιλωτικά προγράμματα και οι δράσεις θα δώσουμε τον λόγο στον κύριο Φερνάντε. Όμως έχει κουβεντούλα τώρα με τον κύριο Μπέγκερ. Μα είπατε, πρόεδρε, ο κύριος Φερναντές, ότι αυτό το συζητούσαμε το απόγευμα. Οπότε και εγώ χαλάρωσα. Αλλά, αφού το συζητάμε τώρα, θα σας τα πω σύντομα. Μιλάμε για 90 πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις που έχουν εγκριθεί. 63 προγράμματα, 27 δράσεις για τη χρήση 16, 39,8 εκατομμύρια, δράσεις 28,1 εκατομμύρια ευρώ και τα προγράμματα είναι μεταξύ 700.000 και 3 δισεκατομμυρίων όσον αφορά τις ε, υποχρεώσεις και 502 εκατομμύρια όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών. Η πρώτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 4 Τρίτου υπευλήθη, η δεύτερη έκθεση της Επιτροπής αναμένεται για... Ελπίζουμε ε, για τότε που θα έχουμε το σχέδιο προπολισμού για το 17. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε συμφωνήσει, αλλά αν υπάρχει κάποιο ερωτηματικό, ευχαρίστω να σας ε, εξηγήσω. Κύριε Γκάιρ, λέει ο πρόεδρος, πώς πάνε τα πράγματα για το 2017. Ακριβώς όπως τα είπε. Κουάζω. Α, μας Μα αν είχαμε και παραπάνω, χρήματα καλά θα ήταν. Γιατί έχουμε πιλωτικά προγράμματα που μπορούν να γίνουν δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ίσως θα πρέπει να δούμε την πρικοδότησή του στο μέτρο του δυνατού. Και να έχουμε υπόψη και τις προθεσμίες για την κατάθεση των προτάσεων, για, τα πιλωτικά, για τις πιλωτικές δράσεις και την υλοποίηση. Ε, ευχαριστώ τον εισηγητή. σας αφήσω όπως πάντα. Ερωτήσεις? Όχι. Λοιπόν, σταματούμε εδώ. Εξετάζουμε το σύνολο των ερωτήσεων. Μας απασχόλησε βέβαια η Τουρκία. Ήταν όμως κρίσιμα τα ζητήματα και πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Ευχαριστώ και συνεχίζουμε στις 3 το απόγευμα.